Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρετε. Παρακαλώ καθίστε. Είχαμε μια ομάδα εργασίας για το Ταμείο Προσαρμογής στην... για την ε, παγκοσμιοποίηση. Και είχαμε και την πρώτη ελληνική περίπτωση που μας απασχόλησε και μία υπόθεση της Ιρλανδίας. Λοιπόν, έχετε την ημερήσια διάταξη, δεν υπάρχουν σχόλια, άρα εγκρίνεται, θεωρώ. Ε, Θα ξέρετε ότι τα σημεία 15 και 16 αντιστρέφονται. Στο 2, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 8ης και 12ης Σεπτεμβρίου. Εγκρίνονται, υπάρχουν σχόλια. Φαίνεται πως όχι, άρα εγκρίνονται τα πρακτικά. Στο σημείο 3, ανακοινώσεις της Προέδρου, ε, θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτή την συνάντηση που όλο ένα και επανέρχεται η οποία, όπως ξέρετε, ακούγεται και στο διαδίκτυο, γι' αυτό να προσέχετε όταν μιλάτε. Με τους συντονιστές είχαμε μία ανταλλαγή απόψεων χτες με τον κύριο Ρισελ, τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και έτσι θα μπορέσουμε να ορίσουμε το πρόγραμμα εργασίας μας για την επόμενη χρονιά λαμβάνοντας υπόψη και τον προγραμματισμό της ίδιας της Επιτροπής. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι μέσα στα πλαίσια της κινητοποίησης του ε, Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχουμε ε, προβλέψει, είχαμε προβλέψει μια συνεδρίαση της Επιτροπής ΠΕΜ όπου ήρθαμε σε επαφή με μία αντιπροσωπεία του συνδικάτου ΣΕΖΕΤΕ και με τα συνδικάτα, συνδικάτα της ΡΕΝΟ για να μιλήσουμε για ορισμένες ε, ε, υποθέσεις που αφορούν το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θα ήθελα να καλωρίσω θερμά την Αλιέντ Καρέ που είναι νέα διοικητική συνάδελφος και ε, νομικός σύμβουλος είναι μαζί μας, είναι εδώ. Παρακαλώ να σας δούμε όλοι. Σας καλωσορίζουμε θερμά. Euh, Η Αλιέτ Κάρε θα αντικαταστήσει τη συνάδελφο και θα μας δώσει ένα οργανόγραμμα έτσι ώστε να ξέρουμε ποιος κάνει τι. Τέλος. Η κυρία Καρή Μαντελή θα είναι στο επίκεντρο της συνεδρίασης, διότι μία ομάδα δημοσιογράφων θα τραβήξει σκηνές. Γι' αυτό να μην ε, φοβηθείτε. Κρίστινσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω τονέζικη μετάφραση, διερμηνία. Να ρωτήσω, έχω παθητικά δανεικά γιατί θα ήθελα να μιλήσω στη συνέχεια σε ένα άλλο σημείο της μερίσιας διάταξης και θα ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα μου. Μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής λιτότητας, λέει πρόεδρος και δεν ολοκληρώνει. Είναι περίεργο γιατί είναι η δεύτερη φορά που έχω γνωμοδότηση και συμβαίνει το ίδιο και πιστεύω ότι πραγματικά είναι προβληματικό αυτό γιατί έχω προτιμάσει την ομιλία μου στα Δανέζικα και δεν ε, μπορώ να την αλλάξω τώρα τελευταία στιγμή. Θα ήθελα να προτείνω με αποσεβασμό προς τον συντάκτη να αλλάξουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη έτσι ώστε να έχουμε διερμηνία προς τα δανέζικα. Διαβάσατε τη σκέψη μου, κύριε Θέρκας. Αυτό ήθελα και εγώ να προτείνω. Να αφήσουμε το θέμα αυτό για αύριο και μέχρι αύριο η μεγάλη ευελιξία αυτού του οίκου θα οδηγήσει σε δραστικές αλλαγές, ε, δηλαδή κάποιος θα θυσιάσει τη γλώσσα του έτσι ώστε να έχουμε τα δανέζικα αύριο. Οι Πορτογάλοι θυσιάζετε τη γλώσσα σας. Όχι, όχι. Κύριε Ντερόζα, τα αγγλικά. Δεν σας πιστεύω. Τα Ιρλανδικά, τα Ιρλανδικά. Κύριε Κρίστενσεν, σας προτείνω να το αφήσουμε για αύριο το θέμα και μέχρι τότε η γραμματεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξευρεθεί μια λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ικανοποιηθείτε αύριο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Ο κύριος Ορή, ουγγρικά έχετε. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά το εξής. Να εκφράσω την ελληνική μου στο συνάδελφο, διότι το θεωρώ απαράδεκτο να μην μπορεί κανείς να εργαστεί στη δικιά του μητρική γλώσσα. Αυτό πρέπει να αποτελεί εγγυημένο αυτό πρέπει να είναι εγγύηση ε, του καθενός ε, ε, ότι θα μπορεί να μιλήσει και να ακούσει τη μητρική του γλώσσα. Θα, πρέπει το, το Σώμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγγυηθεί αυτή την δυνατότητα. Μα εσείς τα έχετε καταφέρει πολύ καλά γιατί έχετε εγκουρικά ακόμα και στους συντονιστές. Έχουμε λοιπόν μία πρόταση που ικανοποιεί το συντάκτη μας, τον εισηγητή, και ίσως θα μπορέσει να προετοιμαστεί για να μας παρουσιάσει το θέμα στα αγγλικά αύριο, εάν σταθεί αναγκαίο. Σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Μπάστος. Πρόεδρε, πάλι λαμβάνω το λόγο στο γλωσσικό γιατί είναι ένα θέμα αρχής. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Έχουμε το δικαίωμα από τη συνθήκη να ζητάμε στις επίσημες συνεδριάσεις να έχουμε τη μητρική μας γλώσσα. Άρα δεν μπορούμε να δεχτούμε σε μία επίσημη συνεδρίαση Επιτροπής του Κοινοβουλίου να γίνονται εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα που είναι ένας χρυσός κανόνας του Ευρωπαϊκού Σχεδίου. Άρα είμαι αλληλέγγυα προς τον δανό συνάδελφο, όπως θα ήμουν αλληλέγγυα και προς οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο, διότι αυτό είναι θέμα αρχής. Θα ήθελα στην Επιτροπή μας να μην γίνεται καμία, να μην ανακύψει καμία παρόμοια κατάσταση, όποιος και να είναι ο λόγος που θα επικαλεστείτε. Δηλαδή, ιδιαίτερα να μην επικαλεστεί κανείς την κατάσταση οικονομικής λιτότητας. Νομίζω ότι όλες ε, οι ομάδες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τον κύριο Κρίστενσεν. Έχουμε μια μικρή αίθουσα η οποία είναι γεμάτη 12 είναι καμπίνες, άρα γίνονται διαιτησίες και δεν μπορεί ο καθένας να έχει τη γλώσσα του, όλοι δηλαδή. Το συζήτησα με την επικεφαλής της γραμματείας και τη στιγμή που υπάρχουν γνωμοδοτήσεις θα πρέπει ο εισηγητής να μπορεί να εκφράζεται στη μητρική του γλώσσα. Κατά τα άλλα, όλοι θα πρέπει να καταβάλουμε μία μικρή προσπάθεια και να κατανοείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις γλώσσες. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας. Επί του ιδίου δεν θα σας δώσω το λόγο, γιατί νομίζω ότι ο καθένας εκφράστηκε επαρκώς. Άλλο θέμα, εντάξει, εντάξει, σας δίνω το λόγο. Thank you, Madam Chair. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Φτώχεια και τον Αποκλεισμό. Έχουμε τις συμβαστικέ μόνο στα γαλλικά. Άρα αυτό αποτελεί πρόβλημα γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο η διερμηνία που αποτελεί πρόβλημα, αποτελεί και η μετάφραση. Τι θα κάνουμε, αύριο έχουμε ψηφοφορία. Μάλιστα, θα το δούμε. Θα το δείξουμε, θα το δούμε, θα το δούμε. Καταρχήν ας ανοίξει το θέμα και ο κύριος Φρεντερίκ Νταρντέν έχει το λόγο για να μιλήσει για τις τροπολογίες στα γαλλικά. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρσι το Σεπτέμβριο αναπέμψαμε το θέμα για λόγους μετάφρασης στα αγγλικά, αλλά αυτό έγινε άτυπα Και αυτό μας επέτρεψε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και να τις ε, συνεχίσουμε υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, έτσι ώστε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό. Μπορέσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε τις εργασίες και νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα συμπέρασμα αρκετά καλό. Δώσαμε δηλαδή τελική μορφή σε ένα μεγάλο μέρος του όγκου εργασίας και με βάση τις 400 τροπολογίες φτάσαμε σε 47 συμβιβασμούς για να φτάσουμε σε σύνολο 200. Νομίζω ότι είναι τροπολογίες συμβιβασμού που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές. Να φτάσουμε δηλαδή σε μία ε, πλειοψηφία. Τώρα, Ως προς τις ε, πιο σημαντικές ε, συζητήσεις, μιλήσαμε για τον ελάχιστο μισθό, για το ελάχιστο εισόδημα, όπου έγινε λόγος για μια οδηγία πλαίσιο, αλλά στο συμβιβασμό η Επιτροπή μίλησε για μια πρωτοβουλία νομοθετικού περιεχομένου, κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό σε σχέση με τις συζητήσεις μας. Υπάρχει και η οδηγία, η οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε ομοφωνία, όμως κράτησε αυτή την πρόταση συμβιβασμού, η οποία είναι αναγκαία. Και ελπίζω να μπορέσει να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Υπάρχει και το SSIG. Εδώ η οδηγία δεν επιτρέπει να φτάσουμε σε συμφωνία. Χρειάστηκε ξαναδούμε κάπως το κείμενο και να επιμείνουμε στο θέμα της ε, προσβασιμότητας ως προς το SSIG. Επίσης, αυτό που μας απασχολεί είναι ο σύνδεσμο μεταξύ οικονομικής διακυβέρνησης και της φτώχειας. Υπάρχει άμεση, άμεσος σύνδεσμος και συνάφεια και μας ενδιέφερε και το πακέτο των έξι νομοθετημάτων καθώς και υπηρεσίες ε, κοινής ωφελίας οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, SSIG. E και δεν αναφερόμαστε άμεσα, αλλά τονίζουμε το γεγονός ότι τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πολιτική απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Αυτό ακριβώς είχαμε αναφέρει και στα πλαίσια αυτής της μνήας. Αυτά είναι ορισμένα θέματα τα οποία μας ε, επέτρεψαν να φτάσουμε σε συμφωνία και να μην παλινοδίσουμε σε σχέση με ειδικά κείμενα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά σημαντικά θέματα, αυτά τα σημαντικά θέματα. Θα πρέπει να γίνουν με ορισμένες μικροπροσαρμογές. Θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τα θέματα αυτά με τη γραμματεία έτσι ώστε να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο και θα ήθελα απλώς ε, και πάλι να πω ότι ευχαριστώ τους μεν και τους δε για τη συνεισφορά τους και για την επικοδομητική τους στάση. Νομίζω ότι στα πλαίσια της παρούσας κρίσης θα πρέπει να εγκρίνουμε μία έκθεση από την Επιτροπή στην Επιτροπή αύριο με βάση την πλατφόρμα στην Κρακοβία λίγες μέρες μετά. Και ελπίζω να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόπες. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας. Ε, καταφέραμε να μιλήσουμε αρκετά επί του εξή θέματος. Ε, μετά από τις 400 αρχικές τροπολογίες φτάσαμε σε 47 τροπολογίες συμβιβασμού και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να εγκριθούν, ανώφιστο στο σύνολό τους, εν Και θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έκθεση και για την σύνοδο της ε, Κρακοβίας. Στην 333, τροπολογία 333, θα ήθελα ξεχωριστή ψηφοφορία είναι η ε, τροπολογία της κυρίας Ντελή που μιλά με το «recommande la mise en œuvre du réglementation». Συστήνει τη θέση σε ισχύ της σύστασης. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με μία ενδεχόμενη επαναδιατύπωση για να μπορέσουμε ενδεχομένως να την υπερψηφίσουμε. Υπάρχει μία τροπολογία, η 368 του κυρίου Τόμας Μαν, η οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο W, στο συμβασμό W. Και επίσης μία άλλη τροπολογία αφορά τα έχοντας υπόψη το όμικρον, το σημείο όμικρον. Είναι η 382. Θα πρέπει να κάνω μαθήματα πολωνικών για να μπορέσω να προφέρω το όνομα της συντάκτριας. Σε σχέση με τα αμαία και πιστεύω ότι η τροπολογία συμβιβασμού όμικρον θα μπορούσε να μας βρει σύμφωνους για να καλυφθεί αυτό το θέμα. Άρα αύριο θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς η Λίν δεν μπορεί να είναι εδώ, οπότε θα ήθελα εγώ να σας παρουσιάσω μερικές σκέψεις της. Η κυρία Λίν θα ήθελα να ευχαριστήσει καταρχάς τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία και για την συνεργασία του με τους κοιόδης εισηγητές. Η έκθεση αυτή είναι περισσότερο αναγκαία σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Και οι σκιώδεις ε, ε, οι συγητές ε, μπόρεσαν να συμβαστούν σε αρκετέ ε, τροπολογίες, όμως, σε αρκετού συμβιβασμού, όμως υπάρχουν άλλε συμβιβαστικές προτάσεις τις οποίες η εισηγήτρια δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει και αφορούν νομοθετικά μέτρα προσβασιμότητα και ελάχιστο εισόδημα. Ε, καταλήγοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την, ε, τον εισηγητή για όλη την ε, καλή του εργασία και ελπίζω να προχωρήσουμε μαλά όλοι αύριο στην ψηφοφορία. Κυρία... Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Έχω μια γενική παρατήρηση Θα ήθελα να αναφερθεί ε, στο προήμιο το θέμα των Ρωμά, διότι όλοι συμφωνούμε ότι ε, αυτή η ομάδα των Ρωμά υποφέρει ιδιαίτερα από κοινωνικό αποκλεισμό. Πιστεύω ότι πρέπει να, να περιληφθεί αυτή η αλήθεια, αυτό το γεγονός και στις συμβαστικές τροπολογίες. Η κυρία Τελίπη μετά η κυρία Κωστά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την εξαιρετική αυτή εργασία. Πολλές τροπολογίες αλλά και πολλοί συμβιβασμοί που μας οδηγούν σε συγκεκριμένες προτάσεις γενικότερου προσανατολισμού και που αντικατοπτρίζουν τη θέση του Κοινοβουλίου εν ώψη της συνεδρίασης της Κρακοβίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τιμήσουμε τα πρώτα θύματα της φτώχειας, είτε είναι οι νέοι, είτε οι γυναίκες, είτε τα άτομα με αναπηρίες και υπάρχει και αυτό το θέμα της κοινωνικής ένταξης που για μένα είναι ύψης της σημασίας. Επίσης, θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της διασφάλισης ειδών διατροφής, της διατροφικής ασφάλειας, θέματα στέγης, εκπαίδευσης, υγείας, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να διάγουν μία αξιοπρεπή ζωή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και η καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων. και μας ενδιαφέρει γενικότερα η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουμε να διανύσουμε ακόμα πολύ δρόμο. Η κυρία Κώστα και μετά ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα την έκθεση διότι μιλά για βασικά θέματα και εγώ από την Επιτροπή Πολιτισμού θεωρώ ότι τα τρία βασικά θέματα λαμβάνονται υπόψη επαρκώς. Μας ενδιαφέρουν και οι εθνικές μεταρρυθμίσεις και μία μείωση της εγκατάλειψης του σχολείου, έτσι ώστε να δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία και στα παιδιά. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο έχει μείνει πίσω η Ευρώπη επί του θέματος. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής κατάρτιση για αυτούς που έχουν εργαστεί και για αυτούς που επιθυμούν να έχουν συνεχή κατάρτιση ή διαβίου κατάρτιση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πολύ μεγάλη εργασία ως προς το ΕΚΤ και τα άλλα ταμεία. Επίσης, ελέγχθη και ίσως θα πρέπει να επαναληφθεί ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιες ανάγκες έχουν οι μειονεκτούντες έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους εντάξουμε πιο στοχοθετημένα. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω για την εισήγηση αυτή. Ο κύριος Τόμας Μαν και μετά η κυρία εδώ. Ο κύριος Τόμας Μαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Φρεντερίκ για τη δουλειά του, αλλά και για τις τροπολογίες που ήταν πολύ άριθμες και πώς τις αντιμετώπισε, κοιτώντα ε, με κριτική διάθεση, αν θέλετε, την όλη διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που δεν διακηρύσουν κάποια ιδεολογία, αλλά ασχολούνται με κάποια συγκεκριμένα θέματα και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει ότι αυτό που απαιτούν πολλοί πολίτες, πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό γιατί και στις τροπολογίες διαπιστώσαμε ότι κατατέθηκαν τροπολογίες από βουλευτές του Κοινοβουλίου μας οι οποίοι προέρχονται από διάφορες ομάδες. Δηλαδή υπάρχει διακομματικά, ε, διακομματικές τροπολογίες. Αυτό δεν το ζούμε σε πολλές εκθέσεις και νομίζω ότι αποτελεί μια σημαντική πρόοδο. Ερωτώ, Φρεντερικ, πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία θα υπάρξει έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία όμως έχει πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να παρουσιαστεί στο Στρασβούργο. Ποια είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος λοιπόν που μπορεί να υπάρξει αυτή η σημαντική δουλειά με τη μεγάλη ηλικία, με τους πολλούς συμβιβασμού που επιτεύχθησαν, με τις ε, πολλές τροπολογίες, με την καλή επικοινωνία. Τι θα απομείνει από όλα αυτά. τι μπορεί να προκύψει από τη δουλειά αυτή. Διαπιστώνοντας ότι σε πολλές από τις χώρες μας δεν κοιτάμε καν το θέμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Και πολλοί λένε ότι α, εμείς προτιμάμε να τα κάνουμε όλα σε εθνικό επίπεδο. Τι σημαίνει λοιπόν μια τέτοια έκθεση, τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα, πώς μπορεί να επιτευχθεί πιο πολύ η Ευρώπη αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ συνάδελφοι και νομίζω... Η κυρία Ιρέδο και μετά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Δίνοντας συνέχεια σε αυτά που είπε ο κύριος Τόμας Μαν, θα ήθελα να τους δώσω μία απάντηση. Πολλές φορές προσπαθήσαμε να εγκρίνουμε κάτι σε σχέση με τους ελάχιστους εθνικούς μισθούς, με το ελάχιστο εθνικό μισθό και να φτάσουμε σε ένα 60% μέσο όρο με βάση κάθε κράτος μέλος. Έμπρακτα ήταν πολύ καλό μέτρο για να μειώσουμε τη φτώχεια και για να κινηθούμε προς την κοινωνική ένταξη. Και θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει. Ε, πρόκειται για μία θέση στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος Φρεντερίκ και νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως να προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα. Πρόκειται όμως για μία συζήτηση η οποία θα διαρκέσει και δεν θα ε, επιληθεί εντάχει. Είχαμε πολλή εργασία, αλλά δεν αρκεί να συμφωνούμε σε διαπιστώσεις περιφτώχειας. Θα πρέπει να φτάσουμε πιο μακριά, να δούμε δηλαδή ποια θα είναι τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν, τα επιμέρους θέματα, ως προς τις πολιτικές που επιδεινώνουν την φτώχεια. Και εδώ ο συμβιβασμός είναι πιο αδύναμος. διότι και ο Φρεντερίκ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές αποδυναμώνουμε το κείμενο. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, η φτώχεια αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς στις χώρες μας μέσα στα πλαίσια των εθνικών πολιτικών ε, λιτότητας. Δεν πρόκειται μόνο για την Πορτογαλία και η κατάσταση θα επιδεινωθεί όσο καλοί και να είναι οι εισηγητέ μας, εάν δεν αλλάξουν αυτές οι πολιτικές και αν παραμείνουν αυτά τα προγράμματα λιτότητας. Θα επιδεινωθεί η κατάσταση και θα πρέπει να αντιπαλέψουμε και με αυτή την ε, βασική αντίφαση, έτσι ώστε να καταγγείλουμε αυτή την κατάσταση ε, υπογραμμίσαμε την θετική εργασία που έχει γίνει, αλλά δεν μπορώ να μην σας διαβιβάσω, ανακοινώσω αυτή τη σκέψη μου. Γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα για να μειώσουμε τη φτώχεια. Κύριε Εάν ε, θέλετε να καταλήξετε να ολοκληρώσετε αυτή την ανταλλαγή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ικανοποίηση που υπάρχει σε σχέση με το κείμενο και το συμβιβασμό στον οποίο μπορέσαμε να καταλήξουμε και μάλιστα εκ μέρους των διαφόρων πολιτικών ομάδων και των συναδέλφων που εκφράστηκαν. Και θα ήθελα να προσπαθήσω, όπως ε, είπα προηγουμένως, να σωματώσω τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν. Αλλά βεβαίως δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί εκ βάθρων αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί μέχρι τώρα. Σε σχέση με τις ε, τελευταίες παρεμβάσεις, θα ήθελα να πω τα εξής. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας θα πρέπει προφανώς να, να έχει τη χρησιμότητά της στο μέλλον και όχι να περιοριστεί στην ε, μικρή συζήτηση η οποία θα λάβει χώρα προσεχώς στο Στρασβούργο. Θεωρώ ότι θα πρέπει καταρχήν να, κατά τη διάρκεια της, συμβασίας, της σύμβασης στην Κρακοβία να επηρεάσει την Επιτροπή και τις χώρες ε, μέλη όσον αφορά διάφορα θέματα, όχι μόνο για να τις ευαισθητοποιήσει, αλλά προκειμένου να υπάρξει και μία πρόοδο σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να υπάρχει μία συνέχεια. Μία συνέχεια ετήσια, εν πάση περιπτώσει, σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο της πλατφόρμας, αλλά επίσης και στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας εδώ. Και πιστεύω ότι το κείμενο αυτό το οποίο είναι το αποτέλεσμα των ε, προβληματισμών όλων μας θα πρέπει να είναι ένα κείμενο αναφοράς τροποτινά, τροποτινά ούτως ώστε ε, να μπορέσει να οφήσει τον Επίτροπο να δει πώς μπορεί να υλοποιηθεί το κείμενο αυτό. Και όπως αναφέρθηκε ήδη από την κυρία Φιγερέδο, υπάρχουν κάποια μικρά βήματα, κάποιες πρόοδοι που ενδεχομένω φαίνονται περιορισμένες ίσως οι μικρές, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι, αποτελούν κάποια βήματα προς άλλες πρόοδους και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να υπάρξει μια συνέχεια αυτή της έκθεσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την έκθεσή σας αύριο, αν δεν απατώμε. Ωραία λοιπόν και θα περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης όπου δίνω το λόγο στη συνάδελφο Λίζα Γιακονσάρη που ούτως ώστε αναφερθεί στις συμβαστικές τροπολογίες και στην οδηγία προποθέσει εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης. Παρακαλώ, κύριε συντάκτη, έχετε το λόγο. Δυστυχώ δεν έχω κάτι νέο να σα αναφέρω. για την έκθεση του κυρίου Κονφεράτη για τους εποχιακά εργαζόμενους ζητήσαμε να γίνει αναβολή της ε, ψηφοφορίας. Γιατί? Λόγω της Επιτροπής Γιούρη, η οποία θα γνωμοδοτήσει επί της νομικής βάσεως στις 10 του μηνός. Επίσης, περιμένουμε ανταπόκριση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. για το πόσο η οδηγία αυτή σχετίζεται με την οδηγία για τους αποσπασμένους. Άρα, θα θέλαμε να γίνει μια κανονική ανάλυση και να υπάρξει απάντηση και επί της νομικής βάσεως. Λάβαμε μια επιστολή από την Επιτροπή. Η επιστολή όμως είναι στα γαλλικά και θα θέλαμε να εξετάσουμε εντελεχώς την επιστολή σε άλλες γλώσσες. Κάποια ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν εκκρεμή κάποια ζητήματα ως προς την κοινωνική ασφάλεια, ως προς τον ορισμό της απαιτούμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επανεξετάσουμε την πρόταση των πράσινων για το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων και δεξιοτήτων προκειμένου να συμπεριληφθεί και αυτό. Επί του παρόντος όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα ήθελα λοιπόν να είναι σαφές το κείμενο με πολύ φιλική προς το χρήστη έκθεση και από κοινού με τον κύριο Γιακολίνο θα θέλαμε να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και αυτό παρουσιάζει κάποια προβλήματα λοιπόν. Έως τώρα ο κύριος Γιακολίνο έχει αποδείξει ότι χρειαζόμαστε τον ορισμό της μπλε κάρτας για τους ε, εξειδικευμένους εργαζόμενους και για τους εκπαιδευόμενους, αλλά έχουμε ένα θέμα για τον ορισμό των managers ακόμα. Επίσης, εξακολουθεί να παραμένει εκρεμές το ζήτημα του κατά πόσο η οδηγία θα καλύψει την τις οικοδομές. Και έχουμε σχόλια και από πλευράς εργαζομένων και από πλευράς εργοδοτών και οι δύο θεωρούν ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί γιατί ε, δημιουργούνται πιο πολλά προβλήματα από ό,τι επιλύονται. Είναι όμως και θέμα αρχής. Θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο μπορεί να εξαιρεθεί ένα τομέα από μια οδηγία. Αυτό ενδεχομένω να προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον. Θα θέλαμε ε, ωστόσο να πετύχουμε καλούς συμβιβασμούς και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά όπως σας είπα περιμένουμε ακόμα τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ε, αποσπασμένους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς που θέλει να πάρει το λόγο. Δεν βρισκόμαστε ακόμα στο τελικό στάδιο γιατί θα περιμένουμε τη γνωμοδότηση της ε, ΛΥΜΠΕ. Εγώ, σε σχέση με το σημείο που αναφέρατε, ε, κυρία Συγκέτρια, ε, το τελευταίο σημείο της παρέμβασής σας, δεν είμαι ειδική για αυτό το θέμα όπως εσείς, αλλά όταν εξαιρούμε το σύνολο του κλάδου των οικοδομών, της κατασκευής, νομίζω ότι πραγματικά ανοίγει ένα μεγάλο χάσμα όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Και ξέρουμε πως ε, η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι, είναι εκρηκτική σε πολλές χώρες μέλη, ε, ειδικά σε αυτό τον κλάδο. Λοιπόν, διαρωτώ με ε, κατά πόσο δεν έχουμε ακριβώς αναγκαστεί την ενεργεία για τον κλάδο αυτό, τον ελόγο κλάδο. Πριν λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα αυτό της εξαίρεσής τους από το κλάδο, νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε κατά πόσο θα πρέπει πράγματι να ψηφίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Λάμπερτ, έχετε το λόγο. Um, Σας ευχαριστώ και μιλάω εξ ονόματα της Ελίζαμπεθ Σρέντερ, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίαση. Θα θέλαμε να πούμε ότι και εμείς συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τη σχέση με την οδηγία με τους απασπασμένους και θα πρέπει όλα αυτά να διευκρινιστούν γιατί ασφαλώς θα πρέπει να μιλάμε για εργαζόμενους και όχι για υπηρεσίες. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς ότι μιλάμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν είναι ουσιώδες για μας. Επίσης ουσιώδες είναι, είναι να υπάρχει ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων σε όλη την οδηγία προκειμένου να προωθήσουμε καλύτερα πρότυπα και όχι να χρησιμοποιηθεί η νομοθεσία αυτή για να πέσουν τα πρότυπα αυτά κάπου σε κάποιες περιπτώσεις. Και πάλι αυτό μας οδηγεί στο καθεστώς του εργαζόμενου. Και φυσικά έχει πολύ σημαντικό σημείο είναι και η αρχή του χώρου απασχόλησης που καθορίζει τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Να πω και εγώ για τον τομέα των κατασκευών, των οικοδομών, ότι, όπως είπε και η Πρόεδρος, αν δεν το συμπεριλάβουμε, θα μείνει ένα μεγάλο χάσμα στην οδηγία, γιατί μετά θα ανακύψει το ερώτημα του πώς θα αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο κλάδο. Αν αρχίσουμε τώρα και τομεακά εμ, αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, που ήδη υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός, θα έχουμε προβλήματα. Επίσης, Νομίζω θα ανακύψουν ερωτήματα περί του πού θα βάλουμε την διαχωριστική γραμμή. Κάποιος ε, που είναι αρχιτέκτονας είναι ή δεν είναι στον τομέα των κατασκευαστικών των οικοδομών. Εγώ είμαι, ξέρετε, από το Λονδίνο και έχουμε και τα Ολυμπιακά ε, έργα. Ε, νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα με τις διαχωριστικές γραμμές. Αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα των ατόμων, ούτε τα συμφέροντα της συνολικής οικονομίας. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Μάλιστα, η κυρία Εσάγια και μετά η κυρία Χίρς, η κυρία Εσάγια, όμως πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το θέμα αυτό. Δεν θα ήθελα να προβώ σε πολιτικές δηλώσεις, γιατί αυτό θα επαναλάμβανε ως αντίλωσο τον Ιούλιο. Θα ήθελα να καλέσω, να πω μάλλον, ότι θα χρειαστεί μετάφραση, όπως είπε και η Λίζα. Θέλω να πω ότι πριν λάβουμε και την έκθεση της της Επιτροπής ε, Λίμπε μπορούμε να αποφανθούμε. Πέρα από την επιστολή στην οποία αναφέρεται η συγγεντριά μας, είχαμε ζητήσει από τον Επίτροπο την ε, ε, ανακοίνωση σχετικά με τις νομικές μελέτες που επέτρεψαν τη σύσταση της βάσης του συνόλου αυτής της νομοθεσίας. Κάτι όμως το οποίο δεν έγινε. Ο Επίτροπος κάνει μνήα στην επιστολή του, η οποία δεν είναι μεταφρασμένη σε μια από τις ε, πιο σημαντικές γλώσσες. Ε, ξαναζητήσαμε λοιπόν από την υπηρεσία της Επιτροπής τη σχετική κοινοποίηση ε, για τη νομική βάση που θα τεθεί ε, στη διάθεση της εισηγήτριας, κυρία Χίρους και στη συνέχεια ο κύριος ε, Μάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταλαβαίνουμε τους συμβιβασμού, αλλά προέκυψαν και κάποιοι συμβιβασμοί μέσω των τροπολογιών. Το θέμα της, ε, του κατασκευαστικού κλάδου θα πρέπει να το συζητήσουμε εκ νέου. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλές και διαφορετικές οι απόψεις για το θέμα αυτό και ότι υπάρχει και το επιχείρημα να αποκλειστεί ο κλάδος αφετέρου. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και τον αντίκτυπο που θα σήμαινε αυτό. Τι θα σήμαινε. Έχουμε τους εξειδικευμένους, έχουμε τους εκπαιδευόμενους. Αυτό μπορεί να ταιριάξει και στον κλάβο τον κατασκευαστικό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα αυτό. Την ιδέα τώρα να γίνει να φορά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων και δεξιότητων δεν την, δεν την βρίσκω κακή. Αλλά αν η κατάταξη είναι τόσο υψηλή που υπάρχει τόσο μικρό περιθώριο ελιγμού, ίσως η οδηγία τελικά να οδηγήσει μην, στο να μην ισχύει για, κανέναν αυτό, αυτή η ρύθμιση άρα είμαι μάλλον επικριτική σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη του πλαισίου αυτού. Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα, για παράδειγμα ε, η, διάρκεια, η χρονική διάρκεια έξι μηνών ή ενός έτους πριν τη μεταφορά. Νομίζω ότι αν τα περιορίσουμε τόσο πολύ και ορίσουμε τόσο λεπτομερώς τέτοιες ε, λεπτομέρειες, θα περιορίσουμε και την χρησιμότητα της οδηγίας αυτής τελικά. Στην έκθεση ε, υπογράμμισα το πιο πολύ Ευρώπη και πάντα αυτό γίνεται πάντα, παρανοείται πάντα. Δεν εννοούμε πιο πολύ κεντρική διαχείριση. Δεν θέλουμε να κάνουμε πιο πολύ γραφειοκρατία, όχι. Εννοούμε από κοινού να βρούμε έξυπνες λύσεις, προκειμένου να ε, ευνοήσουμε τις σωστές εξελίξεις. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε σαφές με την έκθεση αυτή. Θα πρέπει να υπάρξει τέτοια ρύθμιση προκειμένου η ποιότητα των ε, θέσεων εργασίας να μην ε, πέσει, να μην καταστραφούν όσα υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην εντύπωση ότι θέλουμε να αλλάξουμε την κινητικότητα. Όχι, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να έχουμε κριτήρια που να ορίζουν μία βασική ποιότητα, σύμφωνα με τα οποία οι κοινωνικοί εταίροι εξήγαν συμπεράσματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα κράτη-μέλη. Τότε θα έχει νόμιμα η επικουρικότητα και θα είναι σωστή και δεν θα αποτελεί στρατηγική, αν θέλετε, υπεράσπιση εναντίον των άλλων. Και αυτό νομίζω ότι είναι σαφές. Η Jean Lambert μίλησε προηγουμένως για τις διαχωριστικέ γραμμές που θα χρειαζόμαστε. Θα τα χρειαστούμε αν δεν πληρούνται τα κριτήρια. Μία απόφαση λοιπόν για περισσότερη Ευρώπη στην οποία θα συμμετέσχουν και οι άλλες χώρες είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει η ρύθμιση στην οποία θα έχουμε δώσει την απαραίτητη, τον απαραίτητο χρόνο. Γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο κατασκευαστικός κλάδος. Πρόκειται για ένα κλάδο ο οποίος μας έχει απασχολήσει επανελειμμένα στο Κοινοβούλιο και με μεγάλη ε, διαφωνία και Μα είχε πει και τότε ο Επίτροπο ότι δεν επιτρέπεται η υπερβολική ρύθμιση στη γερμανική αγορά γιατί θα καταπνίξει την αγορά. Αντίθετα, εμεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ορίσουμε ποιο είναι ο νόμιμο και ποιο είναι ο παράνομος ε, εργάτη. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει το τι σημαίνει η πιο πολύ Ευρώπη. Όχι ότι το κράτος μέλος θα έχει πλέον ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλειστούν οι κοινωνικοί εταίροι. Ένα ωραίο παράδειγμα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η περισσότερη Ευρώπη ήταν η ομιλία του Μπαρόσο την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο με όλες ε, τις ε, εκφάνσεις της. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έξυπνα επιχειρήματα και να πούμε ότι κοιτάξτε, φυσικά θα συμμετάσχετε και δεν θα υπάρχει κεντρική διοίκηση, κεντρική διαχείριση. Κύριε Μπενάμιν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπατε καθώς και η κυρία Λάμπερτ και ε, όπω και ο κύριο Τόμας Μαν, κάτι που δεν ε, συνηθίζω. Κυρία συγέτρια, λοιπόν, ακούσατε ότι υπάρχει μια πλατιά ε, πλειοψηφία ε, που σας δίνει μια ξεκάθαρη γραμμή όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Δεν νομίζω ότι στη φάση αυτή υπάρχει λόγος να παρέμβετε, ε, εκτός εάν το επιθυμεί. Ναι, θα ήθελα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 θα μιλήσουμε για τους εποχιακά απασχολούμενους με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή υποσχόληση. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αναβληθεί η ψηφοφορία για την Σύνοδο του Νοεμβρίου, αναμένοντας την γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Θα σας δώσω όμως το λόγο για να μας πείτε σχετικά με το επίπεδο της διαπραγμάτευσης και με κάποια κρίσιμα σημεία, επίμαχα σημεία τα οποία δίνουν, ε, θα μπορούσαν να δώσουν λαβή σε κάποια συζήτηση. In attesa appunto del parere della Libe con i giorni che abbiamo guadagnato, stiamo insieme al collega Moro. Ευχαριστώ πολύ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Ε, συνεχίσαμε την προσπάθειά μας να βρούμε ένα συμβιβασμό. Και όσο δυνατόν πλατύτερο ε, συμβιβασμό. Θα ήταν ε, για μας ε, καλύτερο να γίνει αυτή η εργασία από κοινού, ούτως ώστε να προσθεθούν τα πράγματα. Είναι δύσκολο να αναζητεί κανείς κάποιους συμβιβασμούς, αλλά από την άλλη θέλουμε να το διευκρινίσουμε ε, για όλους τους συμμετέχοντες που βρίσκονται τα κρίσιμα σημεία, τα προβλήματα. Και θα θέλαμε να βρούμε ε, κάποιες δυνατότητες να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Τα ερωτήματα τα οποία τα πιο, τα θέματα τα είναι τα πιο επίμαχα, καταρχήν είναι το πεδίο εφαρμογής. Εδώ υπάρχουν πολλές τροπολογίες και οι συνάδελφοι που βλέπουν εδώ κάποια προβλήματα ε, θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ρύθμιση η οποία να αφορά μόνο τους εποχιακά απασχολούμενους. Ε, πρόκειται για εποχιακά απασχολούμενους τον οποίο η εργασία περιορίζεται χρονικά. Ωστόσο αυτό δεν σχετίζεται, δεν συνδέεται άμεσα με την εποχιακή απασχόληση. come capita in più di una εδώ είναι για παράδειγμα ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επετελούν κάποια δεδομένη εργασία σε κάποια, για κάποια χρονική περίοδο χωρίς αυτό να σχετίζεται με τις εποχές του έτους. Επίσης υπάρχουν και άλλα σημαντικά προβλήματα. Πρέπει να γνωρίζουμε ε, για ποιο τομέα μιλούμε και συμφωνούμε για τους τρεις τομείς, τα, τη γεωργία, τα οποροκυπευτικά και τον τουρισμό και διερωτώμεθα πόσο μπορούμε να διατηρήσουμε κάποιο περιθώριο ελιγμών αφήνοντας το, τη δυνατότητα επιλογής να εντοπίσουν χώρες μέλη και κάποιους άλλους τομείς, αλλά υπό την προπόθεση ότι συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή της επιλογής και οι κοινωνικοί εταίροι. Ναι, δεν έχουν το δικαίωμα σχης βέτο, αλλά παρόλα αυτά συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτή την αναζήτηση μιας επιπλέον λύσης εκεί που κάτι τέτοιο θεωρείται αναγκαίο παράλληλα με κάποιες ε, λύσεις που απορρέουν από την οδηγία. Όσον αφορά τη διάρκεια, και εδώ υπάρχει μία σύγκληση όσον αφορά αυτή τη διάρκεια των έξι μηνών. Αλλά αυτοί οι έξι μήνες ε, δεν ε, αφορούν τον ετήσιο κύκλο των 12 μηνών αλλά αφορούν το διάστημα των 12 μηνών και αυτό μας δίνει κάποια ευελιξία σε σχέση με τον τουρισμό επί παραδείγματι. Και κάτι τέτοιο θα έπρεπε να μας επιτρέψει να μην ασκήσουμε κάποιες ε, διαστρεβλώσεις. Κάτι άλλο σημαντικό είναι να, για τη αυτή να επικυρώσουμε την αρχή ισότητα εργασίας, ίση μεταχείριση. Και αυτό ισχύει για όλα όσα ισχύουν με τις, ε, για τις λεγόμενες συλλογικέ ε, συμβάσεις. Η περιγραφή αυτών των συμβάσεων βεβαίω δεν είναι εύκολη γιατί κάθε χώρα έχει τη δική της ε, κατανόηση τη δική της πρακτική για τις συλλογικέ συμβάσεις. Υπάρχουν σε ορισμένε χώρες μόνο εθνικές συμβάσεις, τόπο εργασίε κλπ όπως και να έχουν τα πράγματα, ένα τμήμα αυτής της ε, ίσης μεταχείρισης για ίση εργασία θα πρέπει να τη κατοχυρωθεί μέσω ακριβώ της εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και κατά τα άλλα μέσω της ε, κοινωνικής ασφάλειας η οποία υφίσταται έστω και αν δεν είναι ομοιόμορφη ε, σε όλη την επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους έξι μήνες εποχιακής εργασίας που θα μπορούσε να ενδιαφέρει κάποιον ο οποίο ε, προέρχεται από μια άλλη γωνιά του κόσμου. Κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών, οι εργαζόμενοι αυτών των χωρών και οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα πρέπει να υποφελούνται ακριβώς από τις, ίδιες, ε, από τις ίσες προϋποθέσεις, ή ε, εργασίες από τις κοινωνικές προϋποθέσεις, προϋποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης και από τις συλλογικές συμβάσεις. Και αυτή η βασική προϋπόθεση είναι καθοριστή και αυτό για δύο λόγους. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει ίση μεταχείριση, ή αντιμετώπιση, θα βρεθούμε ενώπιον φαινομένων τα οποία θα αυξήσουν το κοινωνικό dumping. Και από την άλλη υπάρχει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων, οι οποίες ε, θα ε, ε, αλλάξουν την πολιτική Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, ασχολήθηκαν με αυτές τις τροπολογίες. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ καλή βούληση και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση. Κυρία Τουρινέν. Yeah, uh, thanks a lot to the Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε συμφωνία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά φυσικά χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις για το συμβιβασμό που καταρτίστηκε για την απασχόληση. Νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα σας ζητούσαμε να τονίσετε περαιτέρω τον, ε, το θέμα της κοινωνικής ασφάλειας. Να τονίσω ότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό. Καταρχάς ότι τα δικαιώματα μπορούν να εξαχθούν. Δηλαδή, αν κάποιος έχει συνταξιδοτικά για παράδειγμα δικαιώματα, θα πρέπει να, να υπάρχει μηχανισμός προκειμένου να μεταφερθούν στην πατρίδα του τα δικαιώματα αυτά. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος, να έρχεται κάποιος διαρκώς ε, για εποχιακή εργασία στην Ευρώπη. Μιλάμε για χρόνια δηλαδή συνολικά, τα οποία δεν θα έπρεπε να χαθούν τα σχετικά συνταξιβετικά δικαιώματα και σε ό,τι αφορά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Κατά δεύτερον, θα θέλαμε να προσθεθούν και τα δικαιώματα για διακοπές και επίσης το άρθρο 16, κατά τρίτον, θα πρέπει να γράφουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση με τους εθνικούς εργαζόμενους, τουλάχιστον but not limited to, δηλαδή χωρίς να περιοριζόμαστε σε. Αυτό σας φαίνεται ίσως ε, κάπως υπερβελικό, αλλά έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν ότι οι οδηγίες που ορίζουν τα ελάχιστα πρότυπα πολλές φορές από το ΔΕΚ ερμηνεύονται ως τα ανώτατα όρια. Μιλώ φυσικά για την οδηγία για τους αποσπασμένους. Αυτό και απολυτικός αλλά και για νομικούς λόγους, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ερμηνευτεί ως ε, ελάχιστο πρότυπο. Ελπίζουμε τέλος να υπάρξει ένα δυναμικό κείμενο που να αντιμετωπίσει την κατάσταση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει έντονη εκμετάλλευση στους εποχιαρκά εργοζόμενους, οι οποίοι συχνά δεν είναι καν γραμμένοι. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματά τους. Και αυτό θα κάνουμε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και σε ό,τι αφορά την και τις κυρώσεις. Ευχαριστώ Τόμας Χάντελ και Ζαν Λουίκ Μπενιαμίζη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επισημάνω δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο διαπίστωσα και στις δύο εκθέσεις είναι το γεγονό ότι πιστεύω αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια συνέπεια όσον αφορά τον ορισμό ποιο ρόλο παίζουν κατ' ουσία οι κοινωνικοί εταίροι σε σχέση με αυτές τις εκθέσεις. Στην προηγούμενη έκθεση συζητήσαμε κατά πόσο ε, ευθύ εξ αρχή μπορεί να είναι ένα κλάδο, για παράδειγμα ο κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίο επιθυμεί να εξαιρεθεί, έστω και αν συντρέχουν από χρόνε λόγοι. Ε, και έχω κάποιε αμφιβολίε κατά πόσο ε, έχει πολιτικά νόημα να θεσπίζουν κάποιε οδηγίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου τελικά δημιουργείται δεδικασμένο, τετελεσμένο να εξαιρούνται κάποιοι τομείς στους εποχικά εργαζομένους ε, φάνηκε στη σημερινή διαπραγμάτευση για, τις, ε, για τους εμβιβασμούς, όπου το θέμα ήταν κατά πόσο σε εθνικό επίπεδο ε, θα πρέπει να διευρυνθεί το πλαίσιο ρύθμισης πέρα από του τρει τομείς. Αυτό μπορούν να το κάνουν οι κυβερνήσεις μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικού εταίρους. Αλλά αν το ζητούμενο είναι σε εθνικό επίπεδο, μόνο τότε να δοθεί στου κοινωνικού εταίρους το δικαίωμα να αποφασίσουν ε, κατά πόσα θέλουν να συμπεριληφθούν ή όχι, τότε ε, στην περίπτωση αυτή ο κοινωνικός διάλογος χάνει απολύτως την αξία του. Δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι τελικά δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, το έχουν μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θεωρώ ότι αυτό είναι συνεπές αγαπητοί συνάδελφοι και νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να πετύχουμε μια συνεννόηση επί του θέματος αυτό. Ε, ε, κατά πόσο εμείς ε, θέλουμε να δώσουμε στους κοινωνικούς εταίρους όχι μόνο αρνητικά αλλά και θετικά τη, δυνατότητα συμπερίληψη σε μια ευρωπαϊκή, συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Ε, ή να πούμε απλώς ότι ναι μεν έχουν λόγο, αλλά δεν τους παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Δεύτερον, συμφωνώ ρητά με τον συνάδελφο κύριο Κοφεράτη. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ για να εργαστούν, να μην ε, έχουν χειρότερες προϋποθέσεις εργασίας, ε, λιγότερα δικαιώματα, γιατί ε, και θα ήθελα να πόσο πολύ προσεκτικά. Μπορεί κανείς να σχηματίσει την εντύπωση από διάφορες συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτές τις δύο εκθέσεις, ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που έχουν την άποψη ότι αν κάποιοι μαύροι από την Αφρική έρχονται στην Ευρώπη ε, θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι που δουλεύουν εδώ σε καλύτερε προθέσει από ό,τι στη χώρα του. Αλλά κατά τα άλλα δεν θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση με του Ευρωπαίου εργαζόμενου. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη και θεωρώ ότι όλες οι αρχές που διατυπώνουμε στην Ευρώπη και εμπίπτουν στην έννοια ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα κλπ. Ε, εδώ εμπίπτει και το ζήτημα ίση εργασία, ίση μεταχείριση. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτή τη βασική αρχή και θα πρέπει στο πλαίσιο αυτής της επιτροφής να πετύχουμε μια συμφωνία επί του ότι ε, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι, οι πήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να δουλεργάζονται στην Ευρώπη κάτω από ίσες συνθήκες όπως και οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο κύριος Μπεναμιάς, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κάπως θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο χωρίς να μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα για τους ερμηνείς Ωραία. Όλο αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ όλους τους εισηγητές αυτής της Επιτροπής και τους άλλους, γιατί νομίζω ότι προχωράμε πολύ θετικό τρόπο εάν ε, επιτευχθούν αυτοί οι συμβιβασμοί τις επόμενες μέρες. Θα ήθελα να επιμείνω σε ένα τομέα. Είναι ο τομέας που γνωρίζω πολύ καλά, που αφορά μια εξωπρεπή στέγαση όσον αφορά του εποχικά εργαζόμενου στο γεωργικό τομέα, όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, τι αποκαλούμε αξιοπρεπή διαβίωση, αξιοπρεπή στέγαση και εναπόκειται στον ε, εργοδότη να παράσχει μια τέτοια αξιοπρεπή στέγαση. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Άλλοι αναφέρθηκαν στο θέμα της μεταχείρισης, ε, συνθήκες εργασίας ε, και πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση. Νομίζω ότι αν καταλήξουμε σε έναν συμβασμό όπως αυτόν το οποίο επεξεργαζόμαστε για το άρθρο 16 και στο θέμα της μεταχείρισης θα έχουμε επιτελέσει μια εξαίρετη εργασία και αυτή η υπηρεσία πραγματικά θα εκπληρώσει έναν σημαντικό σκοπό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Όμεν Ρόιτερ και στη συνέχεια κυρία Γιάζου Ψιέσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι ζούμε στον Άρη. Ξέροντας ότι για τους εποχιακά εργαζόμενους αλλά και για άλλους υποκόους χωρών έχουμε συμφωνήσει λιγότερα και συμπεριλαμβάνονται λιγότερα στην οδηγία από αυτά που προτείνονται εδώ. Και παρά όλα αυτά, για άτομα τα οποία δουλεύουν μόνο για ένα μικρό διάστημα, όπου υπάρχει μεγάλο γραφειοκρατικό άθος, μπορούμε να πετύχουμε. Θεωρούμε ότι μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά. Μιλάμε για την ίση μεταχείριση εργαζόμενων και αυτό είναι στόχος. Αλλά να ξέρουμε ότι αν τα κλασικά καθήκοντα της κοινωνικής ε, ασφάλειας και εδώ πέρα γίνεται τέτοια αναφορά, αυτό σημαίνει ότι οι εποχιακά εργαζόμενοι θα πρέπει να ασφαλιστούν για όλες τις ασθένειες, είμαι υπέρ, για την ε, μητρότητα, ακόμα και είναι για ατυχήματα, όλα τα οικογενειακά επιδόματα, όλες τις συντάξεις όλα αυτά, όλο την γάμα των κοινωνικών, ε, της κοινωνικής ασφάλειας θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε για άτομα τα οποία εργάζονται για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Φαντάζεστε τι γραφειοκρατικό άχτος συνεπάγεται αυτό. Για τους αποσπασμένους δεν κάνουμε όλα αυτά. Οι αποσπασμένοι ασφαλίζονται στη χώρα από την οποία προέρχονται. Άρα, τι είδους ίση αντιμετώπιση έχουμε υπόψη στο συγκεκριμένο σημείο. Μα πρόεδρε, τα έχω χάσει. Δεν τα καταλαβαίνω πλέον. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ορίσουμε κατά πρώτον ποια περίοδο απασχολείται κανείς ως εποχιακός εργαζόμενος και θα πρέπει να είναι σύντομη. Δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτά που προτείνει το Συμβούλιο και αν υπάρχουν ε, χώρες όπου ο εποχιακός ε, τουρισμός ε, και υπάρχουν επαχιακά εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται κάθε ε, χρόνο και δουλεύουν έξι μήνες, ε, δεν είναι εποχιακά εργαζόμενοι αυτοί. Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε σαν εποχιακά εργαζόμενους. Οι εποχιακά εργαζόμενοι θα πρέπει να διατυπωθούν, να οριστούν με διαφορετικό τρόπο. Αυτοί έρχονται για να μαζέψουν, για παράδειγμα, φράουλες, σπαράγγια. Έχουν άλλου είδους σύμβαση και χρειάζονται άλλου είδους σύμβαση από αυτό που προτείνουμε τώρα και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και δεν είμαστε συνεπείς κοιτώντας όλα όσα συμφωνήσαμε στο παρελθόν. Alors, euh... Κυρία Γεσοφιέσκα και μετά ο κύριος Μπαλτασάρ. Ulega wątpliwości, że wyzwania nie ulega wątpliwości, że wyzwania demograficzne stojące przed Unią Europejską αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε ε, μία σωστή προπαρασκευή αυτής της ε, μετανάστευσης, της υπεύθυνης μετανάστευσης, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ζήσουμε τις ε, αρνητικές απόρριες που σχετίζονται με τα θέματα της ευελίξης ασφάλειας. Θα πρέπει όμως όλοι να έχουν μία αξιοπρεπή εργασία, καλή αμοιβή και σωστή κοινωνική πολιτική. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι εποχικός χαρακτήρας πρέπει να αφορά μία ε, μικρή περίοδο, μία βραχία περίοδο. Και αυτό είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με εκείνους που εργάζονται, που είναι ε, κάτοικοι της χώρας και εργάζονται με εποχικό χαρακτήρα, αλλά ζουν στη χώρα. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποιοι εργάζονται όλο το χρόνο και ποιοι είναι πραγματικά εποχικοί. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να μην συγχαίουμε τους μόνιμους και τους εποχικούς. Θα πρέπει λοιπόν να εισήσει η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να είμαστε ιδιαίτερα συνετοί ως προς την κατανομή όλων των προνομίων και τη χορήγηση των προνομίων. Ο κύριος Μπαλτασάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος υπογραμμίζοντας ένα θέμα, ένα σημείο εκκίνησης. Πρόκειται για έναν ευαίσθητο ε, τομέα όπου έχουμε να κάνουμε με μια δραματική πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι που έρχονται από τρίτες χώρες ε, την χάνουν στιγνής εκμετάλλευσης σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει σύγχυση. Εμείς είμαστε το ΕΛΚ, είμαστε ένα ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα και λαϊκό, το τονίζω αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι οι όροι του 883 θα πρέπει να ισχύουν για τους εργαζόμενους και από χώρες, ακόμα και αν εργάζονται εποχικά. Αυτό είναι το ελάχιστο μετά. Μπορούμε να θέσουμε περιορισμούς ενδεχομένως έτσι ώστε να εξορθολογήσουμε και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Αυτό αφορά και τους Χιώδης και τη Λίμπε, έτσι ώστε να δούμε πώς συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι κατά τη διεύρυνση του τομέα του, των εποχικών, έτσι ώστε να έχουν δικαιώματα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για υποκειμενικό χαρακτήρα, γιατί υπάρχει ας πούμε ένας εργαζόμενος που πάει στα βουνά του Βένετο ή του Τρεντίνο Άλτο γιατί μόνο εκεί μπορεί να εργαστεί θεωρείται εποχικός και ας επανέρχεται κάθε χρόνο. Δεν μας ενδιαφέρει ο επαναληπτικός χαρακτήρας της εργασίας, αλλά η ανάγκη των κρατών μελών να έχουν άλλους εργαζόμενους εκτός από τους μόνιμους. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος επανέλθει πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, η εργασία μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και σκόπιμη. Είχαμε δυσκολίες και κοινά στοιχεία και νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε τροπολογίες συμβιβασμού. Μπορεί να φτάσει ο συνάδελφος ε, Κοφεράτη και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο όπου ο κανόνας είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων από τρίτες χώρες. Είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Η κυρία Χίρς είναι η τελευταία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θεωρώ ότι αυτό το οποίο είναι πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση και υπάρχουν άθλιε συνθήκε εργασία που για μα είναι απαράδεκτε. Και βεβαίω είναι αναγκαίο εδώ να υπάρξουν κάποιε ελάχιστε προδιαγραφέ. Έχω καμιά φορά όμω την εντύπωση, και αυτό αφορά το όσο είπε ο συνάδελφο κ. Χέντελ, ότι δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Δηλαδή θα πρέπει όλα να κινούνται σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα κατάλογο ετοιμάτων, ο οποίο να είναι είναι εφαρμόσιμος ε, και όχι απλώς να λέμε μεγαλό σχήμωνα λόγια, να χτίζουμε παλάτια στην άμμο. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι απαράδεκτο και μεταξύ αυτού που είναι απαράδεκτο και μεταξύ αυτού που ζητάνε ορισμένοι υπάρχει ε, ένα, μια άβυσος. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη χρυσή μέση οδό και γνωρίζω ότι κάποια θέματα όπως η επιμόρφωση για παράδειγμα είναι θέματα τα οποία εδώ θα πήγαιναν υπερβολικά μακριά κατά την άποψή μου ή κάτι που λένε ε, άλλες τροπολογίες, κάποιες περιγραφές σε σχέση με τις συνθήκες στέγασης. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν ε, αποδεκτές, ε, παραδεκτές κατοικίες, αλλά κατά πώς θα πρέπει να είναι τόσο τέλεια η υποδομή, δεν ξέρω. Γιατί ε, αν ε, δουλεύει κανείς στην Ήπεθρο, εκεί οι υποδομές είναι χειρότερες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παραβλέπουμε την πραγματικότητα. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κάποια ρεαλιστικά αιτήματα για ανθρώπους που εργάζονται για μερικές εβδομάδες σε μια περιοχή. Ε, καταλαβαίνω τις επιθυμίες αυτές, τους απότερους στόχους, αλλά θεωρώ ότι τα αιτήματα θα πρέπει να έχουν μια ρεαλιστική βάση. Τελικά και για το λόγο που ισχύει, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να υποφεληθούν από όλα αυτά. Αλλιώς τελικά θα παρακαμφθεί κατ' ουσία η οδηγία αυτή και δεν θα χρησιμεύσει σε απολύτως κανέναν. Κύριε Ισηγητά, θέλετε να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους καταρχήν για τα σχόλια και τις υποδείξεις και θα ήθελα να πω δύο πράγματα επί της ουσίας. Καταρχήν δεν πρέπει να χάνουμε τον απότερο στόχο που μας απασχολεί. Θα πρέπει να ορίσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να αναβαθμίζουν τον εποχικό εργαζόμενο, τον, αυτόν που προέρχεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα πρέπει να το δούμε. Όχι δηλαδή ε, σε σχέση με τον εποχικό και τον εργαζόμενο του χρόνου. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι αυτοί οι εργαζόμενοι να προέρχονται από τρίτες χώρες, να δούμε κατά πόσο προέρχονται από τρίτες χώρες και να τους διέπει το ίδιο συμβατικό δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν η προστασία να είναι η ίδια με τους διαμένοντες. Το θέμα της πρόνοιας θα μπορούσε ε, ενδεχομένως να λυθεί. Δηλαδή ένας εργοζόμενος που έρχεται να εργαστεί θα πρέπει να μπορεί τις εισφορές που έχει καταβάλει να τις πάρει μαζί του όταν φύγει στη χώρα του. Διαφορετικά δεν τηρούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους επανέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ευρώπη, διότι αυτό είναι και ο εποχικός χαρακτήρας, ε, δηλαδή έρχονται, επιστρέφουν στην πατρίδα τους και μετά επανέρχονται. Επειδή υπάρχει ο φόβος να βρεθούν λύσεις που στην ουσία προβάλλουν νέες τυπολογίες, αυτό που έχει σημασία είναι να τονίσουμε τον εποχικό χαρακτήρα. Και νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για εγγυήσεις ίδιων όρων και στους μεν και τους δε. Ως προς ε, τους, ε, τα κοινωνικά συμβαλόμενα μέρη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι κυρίαρχα. Αλλά αν έχει νόημα ο κοινωνικός διάλογος σε τέτοια θέματα, καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση, αλλά δεν σημαίνει ότι θέτουμε στο περιθώριο αυτή τη διάσταση. Γιατί τη στιγμή που συμμεριζόμαστε θέματα αρχής θα πρέπει και οι προδιαγραφές να αντιστοιχούν στις αρχές αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε, λέει η Πρόεδρος, στις 23 Νοεμβρίου και μέχρι τότε θα συμφωνήσουμε, αφού μας γνωστοποιήσει η Λίμπε τη θέση της, θα συμφωνήσουμε. Σημείο 7. Ρενιέ. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για μία αναδιατύπωση. Έχετε το λόγο ως συντάκτρια, κυρία Ρενιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Βρυξέλλες 1 το θέμα μάλλον ήταν μια πολύ καλή και επιτυχής ε, νομοθεσία, ένας κανονισμός. Πρόκειται λοιπόν ένα παράδειγμα το οποίο καταδεικνύει την ε, πρόσθετη αξία της ευρωπαϊκής δράσης. Μετά λοιπόν ε, τη συλλογή εμπειριών έχει έρθει ο χρόνος να γίνει η αναδιατύπωση στο Βρυξέλλες 1 για να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον. Και αναλόγως λοιπόν, αντίστοιχα, η γνωμοτότηση επικεντρώνεται στην ε, Επιτροπή μας στην αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την δικαιοδοσία για τις εργατικές κινητοποιήσεις. Όπως σας είπα, πρόκειται για αναδιατύπωση. Αυτό σας το είπα και την προηγούμενη φορά με λυπή. Λυπάμαι που δεν πρόκειται για πραγματική αναθεώρηση και απλά για αναδιατύπωση. Θεωρώ ότι θα χρειαζόταν αναθεώρηση. Θα επικεντρωθώ στο πόσο στα πρακτικά, στους πρακτικούς ε, κανόνες σε ό,τι αφορά τις εργατικές κινητοποιήσεις. Και το θέμα λοιπόν είναι ποιο δικαστήριο ποια χώρα είναι αρμόδιο, έχει δικαιοδοσία. Σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει να είναι η χώρα εκείνη όπου έλαβαν χώρα εργατικές κινητοποιήσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει αρκετή συνέπεια με τον Ρωμή 2. Επειδή πρόκειται για διατύπωση, θα πρέπει να περιοριστούμε σε ένα στενό πλαίσιο. Δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο. Ο συνάδελφος Μπαλτασάρ στην προηγούμενη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και νομικά αδύνατο να γίνει αυτό που θα ήταν σωστό και ορθό. Να βρεθεί χώρος στον κανονισμό για τον ορισμό του συστήματος. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει η εισαγωγή ενός νέου κεφαλαίου, κατά πάσα πιθανότητα θα αποσύρω την σχετική τροπολογία που αναφέρεται ακριβώς στο θέμα αυτό. Και ανταυτού στο άρθρο 22 θα την τοποθετήσω την πρόταση αυτή. Είναι κρίμα ωστόσο γιατί θα έπρεπε να προσθεθεί ένα κεφάλαιο τέτοιο. Αλλά αυτό νομικός πώς δεν είναι δυνατόν όπως σας είπα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να αναφερθεί στο σωστό σημείο το σύστημα αυτό. Στις τροπολογίες που κατατέθηκαν, ανυπομονώ να δω τις ε, επεξηγήσεις του συναδέλφου Για παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι χρήσιμες ε, οι τροπολογίες αυτές και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το εκλογικό δικαίωμα των εργαζομένων. Θα ήθελα όμως διευκρινήσεις για το άρθρο 19. Και θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις εξηγήσεις των βουλευτών για τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παλτασάρ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα ήταν σκοπιμότερο να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση αφού μας πει η γραμματεία κατά πόσο, κατά πόσο είναι παραδεκτές οι τροπολογίες. Εφόσον πρόκειται για αναδιατύπωση, θεωρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των τροπολογιών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Άρα ε, κινδυνεύουμε να συζητάμε επί του μηδενός, δηλαδή τροπολογίες που αύριο θα δούμε ότι είναι ανεφνομικής υποστάσεως. Θα έπρεπε λοιπόν να μας πει η γραμματεία κατά πόσο είναι παραδεκτές τροπολογίες ή όχι. Κατά την ταπεινότατη μου γνώμη πολλές δεν είναι. Δύο μόνο είναι παραδεκτές. Οι εννέα και οι 16. Όλες οι άλλες ε, εισαγάγουν νέα στοιχεία στην οδηγία και δεν είναι σύμβατες με την διαδικασία αναδιατύπωσης. Ίσως αυτό θα μας βοηθούσε έτσι ώστε να ορίσουμε ποιες τροπολογίες μπορούμε να συζητήσουμε παρά να συζητάμε επί όλων και στη συνέχεια να, να δούμε ότι καμία, σχεδόν καμία δεν είναι παραδεκτή. Συμφωνώ, συνάδελφε, αλλά από ό,τι θυμάμαι στην ε, προηγούμενη μας συζήτηση της Επιτροπής, όταν εξετάσαμε τη γνωμοδότηση, σταθήκαμε επί μακρόν επί το θέμα τους και είπαμε ότι είναι, πρόκειται για επαναδιατύπωση και άρα όταν υπάρχει επαναδιατύπωση ασχολούμαστε με τα θέματα που ξανανοίγει η Κομισιόν και δύο τροπολογίες είναι απαράδεκτες, η 5 και η 16 ενώ οι άλλες αφορούν το νέο πεδίο που έχει ξανανοίξει η Επιτροπή. Άρα δεν βλέπω πού έγκυται η δυσκολία. Κύριε Πόρτας, ελπίζω να μην θέλετε το λόγο για διαδικαστικά. Ο κύριος Χάντελ και μετά κλείνω τον κατάλογο. Έχετε το λόγο. Die Συνάδελφος μου με παρακάλεσε να δώσω κάποιες εξηγήσεις για τις τροπολογίες μου για το άρθρο 19. Θα το κάνω σε εντομία. Ε, κατ' ουσία, ως ε, γραμματέας ε, συνδεκάτων και νομικός εκπρόσωπος των απασχολούμενων είχα σχετιστεί με, το... με θέματα εργαζομένων που μετακινούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και εμπίπτουν σε διάφορα εργατικά δίκαια. Ήταν εργαζόμενοι που εργαζόντουσαν σε μόνιμη βάση σε κάποια άλλη χώρα, αλλά τελικά υπάγονταν στο γερμανικό δίκαιο. Τώρα, όταν ε, υπάρχουν κάποια, θέματα στο χώρο που εργάζεται κανείς ε, τα δικαιοδοτικά όργανα δεν είχαν την ε, αρμοδιότητα να αποφανθούν. Γι' αυτό έχει νόημα στην ε, οδηγία αυτή να δούμε, τι, να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν ο ίδιος ο εργαζόμενος να επιλέξει το δικαιοδοτικό όργανο το οποίο κατά την άποψή του είναι αρμόδιο επί της ουσίας για την υπόθεσή του. Δηλαδή μπορεί να συμβεί ή να πρόκειται για την εργατική σύμβαση ενός Ιταλού εργαζόμενου στην Ρουμανία, ο οποίος είναι μόνιμα εργαζόμενος και ο οποίος ε, ε, βασίζεται στο Ιταλικό δίκαιο. Αλλά θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ε, να μπορεί να επιλέξει το δικαιωτικό όργανο το οποίο είναι ε, αρμόδιο για να αποφανθεί για την υπόθεσή του. Αυτό ήταν το νόημα αυτής της ε, τροπολογίας. Κυρία Εισηγήτρια, εν συντομία, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Φυσικά σημείωσα αυτά που εσείς είπατε, Πρόεδρε, για το θέμα της αναδιατύπωσης, να τονίσω ότι το ίδιο, την ίδια πρόταση επί του περιεχομένου θα τη βάλω σε άλλο σημείο προκειμένου να τηρήσουμε τα στενά πλαίσια τα οποία μας επιβάλλει η αναδιατύπωση. Άρα θα μπει αλλού αυτή η πρόταση, όχι εκεί που είχα προτείνει στην αρχή. Merci euh, Σας ευχαριστώ. Άρα θα ψηφίσουμε επί των ε, τροπολογιών αύριο. adoption en le 6 octobre. Alors, on vote contre Parce que là, celle-ci. Bien, alors contrairement à ce qui est inscrit sur mes, euh, ma fiche, on... Θα ψηφίσουμε σε 7 Νοεμβρίου, έτσι δεν είναι. Κυρία Χίρς. Άρα δεν είχα πληροφορηθεί σωστό Το 8, στο 8 θα δώσω το λόγο στην κυρία ε, ε, Σιλβάνα Ράπτη για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, γειτονίας. Η κυρία Ράπτη έχει το λόγο ως προς το 9 γιατί έχει αντιστραφεί με το 8. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αυτή η έκθεση ήταν να συζητηθεί τη Δευτέρα που έγινε blackout, ε, μετά πήγε στη Δευτέρα του Στρασβούργου που πάλι δεν μπορούσαμε και να την τώρα εδώ ε, συζητάμε και την έκθεση και τις τροπολογίες που έχουν έρθει στο μεταξύ. Ε, υποβλήθηκαν 66 τροπολογίες, οι οποίες είναι όλες ε, στο πνεύμα του κειμένου που έχω καταθέσει και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε με τους ε, σκιώδεις εισηγητές μια πολύ καλή και παραγωγική συνεργασία και σχετικά γρήγορα. Να τονίσω μερικά σημεία. Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία αντιλαμβάνεστε όλοι ότι έχει τεράστια σημασία για την λεκάνη της Μεσογείου και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας εδώ ως, ε, ως ε, Επιτροπή Απασχόλησης, ε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει, να δοθούν, πρέπει να δοθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης βαρύτητα σε δύο σημεία. Η ευρωπαϊκή πολιτική ε, γειτονίας να στοχεύει σε οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έχοντας δύο σημεία. Πρώτον, την απασχόληση στο επίκεντρο και δεύτερον, την τήρηση των κανόνων εργασίας. Ιδιαίτερα η τήρηση των κανόνων εργασίας είναι βασική προϋπόθεση για να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις. Οι προσπάθειες που γίνονται για δημοκρατικές αλλαγές στα κράτη της Βορείου Αφρικής ε, προήλθαν κυρίως από άτομα νέα σε ηλικία, αλλά ταυτόχρονα προήλθαν και από άτομα που βίωσαν την άμεση κατανομή του πλούτου από ανθρώπους φτωχούς, από ανθρώπους που είναι άνεργοι. Αυτά όλα πρέπει και οφείλουμε να τα λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με τις προτάσεις που θα κάνουμε μέσω της γνωμοδότησής μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, σημειώνω ακόμη ότι η δημιουργία, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία θέσεων εργασίας γιατί θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο της παράνομης ε, μετανάστευσης, κάτι που πλήττει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα τις χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην υπάρξει διαρροή εγκεφάλων από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, γιατί αυτό δεν θα βοηθήσει να αναπτυχθούν εκεί οι οικονομίες και η κοινωνία. Πρέπει να ενισχυθεί τέλος ο κοινωνικός διάλογος. Και κλείνω λέγοντας ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά και να παρακολουθεί στενά τα όσα θα γίνονται εκεί, το, τα όσα τις εξελίξεις που θα υπάρχουν εκεί προκειμένου και να δίνει τις χρηματοδοτήσεις αλλά να τηρούνται και όλα όσα πρέπει σε σχέση με την απασχόληση, ε, σε σχέση με τις παράτυπες και παράνομες μορφές εργασίας, σε σχέση με την τήρηση των κανόνων για αξιοπρεπή εργασία προς όλους. Εδώ βάζω μία τελεία και είμαι πρόθυμη να ακούσω τους σκιώδεις των άλλων ομάδων. Έχω δει ήδη τις τροπολογίες, τις κοιτάζω και τώρα, ήρθαν σήμερα το πρωί. Ε, νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή και αποδοτική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Merci. Euh, Η κυρία Merci, Madame la Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ράπτη, την ε, συντάκτριά μας για την ανάλυση που μας έκανε. Νομίζω ότι πράγματι σε αυτή την ε, πολιτική γειτονία και ιδιαίτερα με τη Βόρεια Αφρική έχουμε να κάνουμε με ένα σημαντικό θέμα που θα πρέπει να κινητοποιηθούμε διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ του επίπεδου, ε, της ποιότητας ζωής και επίπεδου ζωής μεταξύ Νότιας Ευρώπης και Βόρειας Αφρικής. Γι' αυτό το αντιμετωπίζουμε και την παράνομη μετανάστευση και θα πρέπει, την οποία θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ορίζοντας σαφώς προδιαγραφές για τις ενδιαφερόμενες χώρες από όπου υπάρχει μετανάστευση προς την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των ε, γειτόνων χωρών για να υποστηρίξουμε την δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα είχε κανένα νόημα να καταπολεμήσουμε στο διηνεκές μακροχρόνια, δηλαδή την παράνομη μετανάστευση, αν δεν μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την κατάρτιση και την εκπαίδευση στους γείτονες. Θα ήθελε κάποιος άλλος να επέμβει. Φαίνεται πως όχι. Κύριε Ράπτη, θέλετε να λάβετε το λόγο εκ νέου για να ολοκληρώσετε. Ε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Σαρτιέ. Οι τροπολογίες που έχει υποβάλει ε, δείχνουν ε, την τεράστια εμπειρία που έχει στο χώρο του Κοινοβουλίου και την ευχαριστώ γιατί με βοηθάει να γίνομαι και εγώ καλύτερη στη δουλειά μου. Ε, νομίζω ότι θα συνεργαστούμε εξαιρετικά. Εξάλλου συνεργαζόμαστε και στο επόμενο θέμα, στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπου εκείνη είναι ε, η συγγήτρια και ο Γοσκιώδης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ε, θα προχωρήσουμε με βάση το χρονοδιάγραμμα. Parfait. Alors, dans ce cadre-là... Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος adopterons ce projet d'avis. Θα εγκρίνουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης 7 Νοεμβρίου. Και αυτό 7 Νοεμβρίου, λέει η Πρόεδρος. Φτάνουμε τώρα στο 10 της ημερήσιας διάταξης στην ακρόαση. Μία μίνι ακρόαση γύρω από την έκθεση Μόρα για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους που προέρχονται από φυσικούς παράγοντες, ιδιαίτερα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και μιλάμε για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μόρα για να μας κάνει μία εισαγωγή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε σκεφτήκατε να διοργανώσουμε αυτή τη μίνι ακρόαση σε ένα θέμα το οποίο είναι τεχνικής υφής, αλλά επικεντρώνεται στην υγεία των εργαζομένων που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έχουμε να κάνουμε με ένα κείμενο, μια οδηγία του 2004, η εφαρμογή της οποίας μεταφέρθηκε τον Απρίλιο του 2012, διότι όπως είχε προετοιμαστεί δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, καθότι ορισμένοι τομείς δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν με βάση τις αποφάσεις αυτής της οδηγίας. Και ιδιαίτερα ως προς το σύμφωνο της χρήσης ή μη χρήσης της απεικόνησης μαγνητικού συντονισμού. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει ε, οπωσδήποτε μία κινητοποίηση, διότι η μη χρησης της απεικονησης μαγνητικου συντονισμου υπαρχουν λοιπον υπαρχει οπωσδηποτε μια κινητοποιηση διοτι ηλικίας είναι πιο υψηλέ από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτό δεν το εφήβραμε εμεί. Βασιστήκαμε σε αυτά που μα συστήσε η Διεθνή Επιτροπή αυτή. Επίση, έχουμε ένα κατάλογο εργαλείων για να διευκολύνουμε τη ζωή των εργοδοτών. Θεωρήσαμε ότι ένας στάνταρ κατάλογος θα βοηθούσε. Προκειμένου να ψάχνει ο κάθε εργοδότης τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί, κατευθείαν στον κατάλογο αυτό και να ξέρει ποια είναι η έκθεση δεν χρειάζεται πλέον να κάνει μεμονωμένε μετρήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις. Και επίσης ε, στα παρατήματα δίνουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα προστασίας. Επίσης, ε, δώσαμε καλύτερη προσοχή σε ομάδες κινδύνου, για τις έγκυες για παράδειγμα. Άτομα με βηματοδότες που έμεσα επηρεάζονται από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και τώρα να περάσουμε στην τελευταία διαφάνεια. Προβλέψαμε επίσης κάποιες περιορισμένες ε, παρεκκλήσεις. Περιορισμένες λέω, γιατί όπως είπα στην αρχή, ότι όλες οι δραστηριότητες και όλες οι κατηγορίες εργαζομένων καλύπτονται από την οδηγία. Αλλά για κάποιες κατηγορίες ισχύουν διαφορετικά ελαφρώς πράγματα από ό,τι για τις υπόλοιπες. Η πρώτη είναι τα ιατρικά μηχανήματα απεικόνιση τα MRI, όπου θα ισχύουν όλα τα υπόλοιπα εκτός από τις ε, μη δεσμευτικές τιμές έκθεσης. Δώσαμε κάποια δυνατότητα στις αναπλές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουν την διαλειτουργικότητά τους, γιατί ξέρετε ότι 22 μέλη της Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ και επίσης για την βιομηχανία και λοιπούς φορείς προτείναμε, προβλέψαμε μάλλον, μία προσωρινή παρέκκληση για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα σταματήσω όμως εδώ, γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλες εισηγήσει και φυσικά είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους άλλους μας προσκεκλημένους. Καταρχήν, ε, εκπροσωπώντας την Business Europe η κυρία Ρεμπέκα Σμιθ που είναι αρμόδια για κοινωνικά θέματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Απασχόλησης και επίση τον εισηγητή που μας προσεκάλεσε να παρουσιάσουμε τη δική μα θέση για το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να, το συντομότερο δυνατό να κάνω κάποιες παρατηρήσει γενική φύση σε σχέση με το πώ βλέπουμε εμεί την αναθεώρηση τη οδηγία και στη συνέχεια θα αναφερθώ σε ορισμένα ειδικότερα θέματα στην αναφερμένη πρόταση της Επιτροπής. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε ότι η αναθεώρηση της οδηγίας είναι αναγκαία για να εξασφαλίσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορούν όλοι οι τομείς να εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας. Ο σκοπός θα είναι μια προσέγγιση βασισμένη στη μείωση, στην αξιολόγηση του κινδύνου και εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων. Εκεί που τα ηλεκτρομαγνητικά ε, πεδία αποτελούν ένα κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων. Ε, πιστεύουμε ότι η οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί κατά τρόπο που να βρεθεί μια λύση για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ε, χειρίζονται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Επίσης πιστεύουμε ότι η οδηγία θα πρέπει να συμπληρωθεί από κάποιες κατευθυντήριες ε, ε, γραμμές ε, και μια ενημερωτική εκστρατεία ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν καλύτερα τις διατάξεις της οδηγίας. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, πιστεύουμε ότι πραγματικά συνιστά σημαντική βελτίωση προ προς την οδηγία και ελπίζουμε οι βελτιώσεις αυτές θα παραμείνουν όσο προχωράμε σε μαθητική διαδικασία παρόλο που απομένουν ορισμένοι τομεί ενισχύς κατά την άποψή μα. Καταρχήν όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και τους ε, ορισμούς που περιλαμβάνονται στην οδηγία αυτή. Θεωρούμε ότι περιορίζεται στην αντιμετώπιση κινδύνων ε, στις ε, βραχυπρόθεσμες ανεπιθύμητες, στα βραχυπρόθεσμα ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ε, αυτό είχε γίνει αρχικά στην πρόταση 2004 και θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει στην αναθεωρημένη πρόταση. Επίσης πιστεύουμε ότι η νέα πρόταση συνιστά, κάνει μια χρήσιμη διάξη μεταξύ ε, επιβλαβών ε, συνεπειών για την υγεία και επιβλαβών ε, αποτελεσμάτων για την ασφάλεια. Θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση και κατά πόσο υπάρχει μια συνέπεια για την υγεία ή όχι. Ωστόσο, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στους ορισμούς και κατά πόσο θεωρούμε ότι είναι ενδεδεγμένα για την οδηγία. Για παράδειγμα, ε, όσον αφορά τι αναπιθύμητε επιπτώσει για την υγεία, ε, θεωρούμε την ε, γενική ευημερία στον χώρο υγείας. Προβλήματα υγείας επηρεάζονται από πολλούς παραμέτρους και ενδεχομένω θα υπάρξει κάποια σύγχυση για να αναγνωρίσουμε κατά πόσο τα προβλήματα υγείας προέρχονται πράγματι από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το ίδιο ισχύει και με την ε, ναυτία, για παράδειγμα, είναι τη ζάλη, σαν άμεσο αποτέλεσμα τη έκθεση στην ακτινοβολία, γιατί τέτοιου είδου ε, συμπτώματα μπορούν να, να προκληθούν από άλλου παράγοντε. Και δεν υπάρχουν ε, όροι όπω προσωρινή ενόχληση. Για παράδειγμα, Υπάρχουν ε, πώς γνώμη πώς ε, προσωρινή ενόχληση που ενδεχομένω θα προκαλέσει κάποια σύγχυση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα τι οριακές τιμές, έτσι όπως υπογραμμίζονται στην οδηγία, πιστεύουμε ότι, κατα... ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη συμπερίληψη οριακών τιμών που να είναι άμεσα μετρήσιμες. Και πραγματικά θεωρούμε ότι οι οριακές τιμές, οι ΚΝΕΠ, ε, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Και πιστεύουμε ότι αν κάποιες εταιρείες χρησιμοποιούν ε, κάποιες επιστημονικές προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες, όπως για παράδειγμα αυτές που χρησιμοποιούνται σε εθνικό πλαίσιο, θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν. Επίσης πιστεύουμε ότι η δυνατότητα να περάσει κανείς σε κάποια επίπεδα δράσης εφόσον οι εταιρείε αυτές μπορούν να δείξουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις, αυτά τα επίπεδα έκθεσης. Αυτό μπορεί να είναι θετικό. Ωστόσο δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες σε σχέση με το πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ορικές τιμές από τις εταιρείε. και αυτό μπορεί να καταλήξει κάποια σύγχυση, έλλειψη αβεβαιότητας και τελικά σε μια έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας, κάτι που θα είναι επιζήμιο για όλους. Επίσης ε, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες ανεπιθύμητες αρνητικές ε, συνέπειες όταν κάποιες από τις οριακές αυτές τιμές, για παράδειγμα σε διαδικασίες συγκόλλησης, που υπερβαίνουν ορισμένα από τα όρια της οδηγίας, ε, παρόλα αυτά δεν καταλήγουν σε επιζήμια για την υγεία αποτελέσματα. Και υποστηρίζουμε πάρα πολύ τη θέσπιση ε, την εισαγωγή ε, κάποιες ευελιξίες στην ενθερμένη πρόταση της οδηγίας. Γιατί για ορισμένε διαδικασίες, όπως είπα, οι ορικές ε, τιμές δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι στην ενθερμένη οδηγία υπάρχει περιορισμένη ευελιξία στις χώρες ε, μέλη όσον αφορά κάποιες ε, αποκλήσεις για ορισμένε επιχειρήσεις και αυτό βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου υπολεγχόμενες συνθήκες. Αυτή είναι το μη κλειδί για μας και υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία θεωρούμε ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποια σύγχυση, να είναι προβληματικά σημεία στην οδηγία. Δεν θα ήθελα να μπω εδώ σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να φέρω ορισμένε από αυτές. Καταρχήν, οι απαιτήσει ε, για ενδείξει ασφαλείας ή τον περιορισμό πρόσβασης σε ορισμένους ε, τομείς. Πιστεύουμε ότι σε ορισμένες ε, περιπτώσεις οι απαιτήσει σε αυτέ ασφαλίε, ασφαλίε δεν είναι εφαρμοστέ και είναι υπερβολικέ. Επίση, πιστεύουμε ότι η τον περιορισμο προσβαση σε ορισμενου τομει πιστευουμε οτι σε ορισμενες περιπτωσεις οι απαιτησει αυτες ασφαλεια δεν ειναι εφαρμοστε και ειναι υπερβολικε επισης πιστευουμε οτι η οδηγια πλαισιο για την υγεία επαρκώς διατυπώνει τι είναι καθοριστικό για την διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων. Και οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις στην ελόγω οδηγία μπορούν να προκαλέσουν κάποια σύγχυση και σε ορισμένες ε, περιπτώσεις να έρθουν σε αντίθεση με άλλα τμήματα της οδηγίας. Επίσης συμφωνούμε ότι ο κατάλογος του εξοπλισμού που ε, ήδη ε, έχει αναφερθεί είναι εξαιρετικά βοηθητικός για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο θα υπάρξει δυσκολία ο κατάλογος αυτός να ενημερώνεται συνέχεια να είναι πλήρες. Γι' αυτό ίσως θα ήταν προτιμητέο να είναι ένα είδος ε, επιπλέον κειμένο, αλλά μην περιληφθεί ο κατάλογος αυτός στο ίδιο το κείμενο της οδηγίας. Εν κατακλείδη θα λέγαμε ότι υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στην οδηγία και ήμουν ευτυχής ε, κατά τη συνεργασία μου με την Επιτροπή, επίσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Ωστόσο, όπως είπα, υπάρχουν ακόμα ορισμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Ελπίζουμε ότι θα αποφύγουμε την προηγούμενη κατάσταση που ε, ε, και νομίζω ότι όλους μας συμφέρει. Γιατί ε, ε, στην προηγούμενη, η προηγούμενη οδηγία δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί άμεσα. Ε, νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποφευθεί αν υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Τώρα, εκ μέρους των συνδικάτων. Ο κύριος Μάρκ Σαπίρ. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Μάρκ Σαπίρ. Είμαι πρώην υπεύθυνος του Τμήματος Υγεία και Ασφάλεια ασχολήθηκα επι μακρόν με αυτά τα θέματα και γι' αυτό πολλοί συνάδελφοι μου ζήτησαν να είμαι παρόν. Έχω παρακολουθήσει την όλη συζήτηση διαχρονικά ως προς τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πριν μπω στο περιεχόμενο της οδηγίας, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας σε ένα βασικό μήνυμα είμαστε υπέρ αυτής της οδηγίας. Πρέπει να γίνουν ορισμένες αναδιατυπώσεις. Πρόκειται για μια συζήτηση που διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια. Αρχίσαμε στη δεκαετία του 90, στις αρχές. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα οδηγία. Δεν υπάρχει ένα εφαρμοστικό μέτρο. Θα θέλαμε λοιπόν αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να καλύψει την αδράνεια της Επιτροπής Επιθεμάτων θεμάτων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Γιατί είχαμε και την αναθεώρηση οδηγίας για τις καρκινογόνες ουσίες που είναι η πρώτη αιτία θνησιμότητας και περιμένουμε τις προτάσεις αυτές εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό τα ευρωπαϊκά συνδικάτα συμμετείχαν στον κοινωνικό διάλογο και είπαμε ότι ταντσόμαστε υπέρ δεσμευτικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Υπάρχουν όμως ορισμένες επιφυλάξεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερις που είναι μείζονες επιφυλάξεις και γι' αυτό θεωρούμε ότι η οδηγία δεν προστατεύει επαρκώς τους εργαζομένους. Το πρώτο θέμα που αντιτίθεται κάπως στη Business Europe είναι ότι η οδηγία αφορά τις άμεσες συνέπειες των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και δεν μιλά για τις επιπτώσεις, τις ορευτικές επιπτώσεις μακροχρόνια. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2008 ζητούσε από την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτό το μακροχρόνιο χαρακτήρα και η ΙΑΡΚ που ασχολείται με θέματα αντιμετώπισης καρκίνου έκρινε ότι θα έπρεπε να ασχοληθούμε με τα ηλεκτρομαγνητικά παιδεία. Θεωρούμε λοιπόν ότι η έκθεση θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλή. Για μας αυτό το θέμα δεν μπορεί να αναβάλλεται στο δινεκές. Το άλλο θέμα είναι η ιατρική επίβλεψη και εποπτεία. Για μας αυτό το ζήτημα είναι ένα μείζον ζήτημα και θα ήθελα να υπενθυμίσω δύο στοιχεία κάθε επιστημονική επιτροπή της Κομισιόν μιλά για επιπρόσθετα στοιχεία για τους εργαζόμενους που εκτίθενται όλο ένα και περισσότερο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα δεδομένα για να δούμε ποιοι εκτίθενται περισσότερο. Από την άλλη πλευρά σας υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο όταν εξέτασε την οδηγία του 2004 συγκεκριμενοποίησε θέματα αρχής της οδηγίας λέγοντας ότι όταν, όταν ξεπερνάμε τις οριακές τιμές ο εργαζόμενος θα πρέπει να βρίσκεται υπό ιατρικό έλεγχο και εποπτεία. Τώρα βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα σε σχέση με το φάσμα συχνοτήτων έκθεσης, αλλά για μας η αρχή είναι ότι δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση των οριακών τιμών, διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει ιατρική επίβλεψη. Βεβαίως ε, αντιμετωπίζουμε και το εξής θέμα. Δεν θα το θίξουμε εδώ. Μας ενδιαφέρει και η ποιότητα της ιατρικής επίβλεψης. Είναι ένα δύσκολο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τίθεται και το ζήτημα των επαγγελματικών ιατρών. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια πρόσωπα είναι πρόσωπα υψηλού κινδύνου, ποιοι είναι οι εργαζόμενοι υψηλού κινδύνου. Πιστεύουμε επίσης ότι χρειάζεται ιατρική εποπτεία και ο ιατρός θα πρέπει να προβεί στα διαβήματα πληροφόρησης του εργοδότη. Ένα τρίτο ζήτημα που σχετίζεται με τις οριακές τιμές και το φάσμα συχνοτήτων αφορά το εξής. Όλα τα μέτρα αυτά, όλες αυτές οι μετρήσεις αφορούν την πρόληψη στο χώρο εργασίας. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι οριακές τιμές που συνελέγησαν με βάση τη αίτημα της ΙΚΝΕΠ και θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται με τις χαμηλές ε, ε, συχνότητες. γιατί μας ενδιαφέρει να προστατεύουμε την ε, υγεία για το νευρικό περιφερειακό σύστημα, για το νευρικό κεντρικό σύστημα και γι' αυτό μας ενδιαφέρει η μέτρηση το, όλων των συχνοτήτων. Επίσης, οι εργαζόμενοι μετατίθενται ή αλλάζουν χώρο εργασίας. Γι' αυτό θα πρέπει να βλέπουμε διαφορετικές οριακές τιμές ανάλογα με το χώρο εργασίας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κινηθούμε προς τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας. Θα πρέπει να ισχύσει ένα σύστημα υποχρεωτικών οριακών τιμών για να γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση πραγματικά βρίσκεται ο εργαζόμενος. Να μην μιλάμε για υποθέσεις. Ένα τελευταίο θέμα είναι ότι τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ασχολούνται με το θέμα της κάλυψης όλων των εργαζομένων από αυτή την οδηγία. Ως προς την μαγνητική απεικόνηση θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο ε, συνέδραμε ουσιαστικά και το ζήτημα είναι να δούμε ποιες εξαιρέσεις και ποια είναι η φύση των εξαιρέσεων που θα πρέπει να ισχύσει. Αυτό το ζήτημα το αντιμετωπίζεται. Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ανέφεραν ότι αναγνωρίσουν την εξαίρεση για εξοπλισμούς με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, αλλά απαιτούν τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα, έτσι ώστε να μην υπάρχει πληθώρα εξαιρέσεων και να υπάρχουν μέτρα σαφούς προστασίας για τους εργαζόμενους αυτές οι εθνικές αποφάσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Κομισιόν έτσι ώστε να υπάρχει αντίστοιχη κάλυψη των εργαζομένων. Υπάρχουν όμως και άλλες εξαιρέσεις. Δηλαδή αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων. Θεωρούμε ότι το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων θα πρέπει να είναι επαρκώς οριοθετημένο και να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας μέσα στα πλαίσια των τεχνολογικών εξελίσεων, διότι οι τεχνολογίες εξελίσσονται άρδιν και θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο είμαστε ενημερωμένοι ή όχι. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το κείμενο της οδηγίας θα βελτιωθεί έτσι ώστε ο εργαζόμενος να προστατεύεται και να προστατευτεί εν ευθέτω χρόνο και ελπίζουμε και εθνικοί εμπειρογνώμονες να μπορέσουν να συνδράμουν την Επιτροπή με τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανωθούμε καλύτερα ως προς την οδηγία πλαίσιο η οποία θα πρέπει να πλαισιώνεται και από εθνικούς εμπειρογνώμενες. Και θέλουμε να περάσουμε από τη θεωρία στο διατάφτα. Σας ευχαριστώ και ελπίζω το συντομότερο να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η οδηγία. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος παρεμβαίνος ο κύριος Τέρι Ούλμερ. Είστε επικεφαλής του Τμήματος Υγεία και Ασφάλεια στο Συμβούλιο Ευρωπαίων Εργαζομένων. metal uh, engineering based industry. Ε, θα μας ε, πείτε κάποια πράγματα σχέση με τις σχέσεις με το Business Europe. Τι σχέση έχετε με το Business Europe. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την ΣΥΜΕΤ σήμερα στην Επιτροπή σας. Θα βρείτε στη διαφάνεια τα θέματα τα οποία θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τα επόμενα 10 λεπτά. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές θα μειώσω και τις διαφάνειες στις οποίες θα αναφερθώ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όλα τα σχόλια που έκανε ο συνάδελφος από την Business Europe. Η CIMET δεν έχει κάποια σχέση σύνδεση με την Business Europe. Βλέπετε ότι εκπροσωπούμε τα συμφέροντα μεγάλης σειράς ε, οργανώσεων από το τομέα της μεταλλουργίας, της Μηχανογείας και ε, που ασχολείται με θέματα τεχνολογίας. Ως οργάνωση υποστηρίζουμε την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στην ε, ασφάλεια και στην υγεία και συμμετείχαμε σε όλες τις φάσεις την διαμόρφωση της οδηγίας και θέλουμε να διαμορφωθεί με αναλογικό και απλό τρόπο η οδηγία για να είναι εύκολη προς την, ε, προς την εφαρμογή και για τους εργαζόμενους αλλά και για τις αρχές. Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω πρόοδος. Ε, η ΣΥΜΕΤ εξακολουθεί να ανησυχεί ότι κάποια από τα μέτρα που προστατεύουν τους εργαζόμενους ε, ουσιαστικά εμποδίζουν τη δημιουργία και την παραγωγή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές για το διάστημα και τις, ε, για, τις, για τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας εξηγήσω τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Νομίζω ότι ίσως να άξιζε τον κόπο να το κοιτάξουμε για λίγο. Μπορούν να προκύψουν ε, σε φυσικό περιβάλλον, αλλά συχνά έχουμε ανθρωπογενή μη ιονίζουσα ακτινοβολία όταν υπάρχει και χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια. Θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ ιονίζουσας και μη ιονίζουσας. Η ιονίζουσα προφανώς συνδέεται με την πυρηνική ενέργεια και έχει διαφορετικό δυναμικό από ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες. Σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές, μιλάμε για τηλεπικοινωνίες, φούρνη μικροκυμάτων, γενική μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε δύο είδη ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έχουμε υψηλή ισχύω ε, ηλεκτρικά πεδία και έχουμε και τα μαγνητικά πεδία τα οποία χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ροή ηλεκτρικών πεδίων. Και το σημαντικό λοιπόν είναι να ξέρουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος στο ανθρώπινο σώμα για να τα βάλουμε όλα στο σωστό πλαίσιο. Έχουμε συζητήσει ήδη, υπάρχει η αρχή της διάκρισης σε ζώνες, δύο κατηγορίες ουσιαστικά. Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών, κοιτώντας. Ε, τις χαμηλές ε, συχνότητες. Μπορεί να μην υπάρχει κανένας αντίκτυπος, μπορεί να υπάρχει κάποια ε, πρόκληση και αντίκτυπος για τα νεύρα. Κάποια, κάποιος ήλικος, ναυτίες σε ακραίες περιπτώσεις. Με όλα αυτά όμως, ε, με προκαλούν ίσω δυσάρεστη αίσθηση, αλλά με το που κλείνει το ρεύμα, με το που κλείνει, το πεδίο, σταματούν αυτές οι δυσάρεστες ε, παρενέργειε. Σε πιο ύψηλε συχνότητε έχουμε θέρμανση των ιστών και πιο ακραία φαινόμενα, ακόμα και εγκάβματα. βλέποντα λοιπόν ε, τον αντίκτυπο, διαπιστώνουμε ότι πιο υψηλό αντίκτυπο έχει υψηλή συχνότητα. Το ερώτημα για την Επιτροπή εδώ είναι κατά πόσο η οδηγία θα πρέπει να βασίζεται σε μια αρχή πρόληψης. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, οι ε, καζόμενη ο εικαζόμενος, ε, οι καζόμενες βλάβες στην υγεία των εργαζομένων. Το θέμα είναι ποιος είναι υπεύθυνο για να τα αποδείξει αυτό. Ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης. Βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους κινδύνους θεωρούμε ότι θα πρέπει οι σχετικοί κίνδυνοι να ληφθούν υπόψη. Από πλευρά της ΣΥΜΕΤ πρέπει να πούμε ότι θεωρούμε ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται παρκώς ε, στην ε, υφιστάμενη οδηγία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αν εφαρμοστεί η μελλοντική οδηγία θα παρέχει την χρειαζόμενη και αναλογική προστασία. Θα ήθελα να μιλήσω για την αρχική αξιολόγηση της ρύθμισης. Προφανώς έχουμε ήδη καθυστερήσει να το ξανασυζητήσουμε αυτό γιατί η αρχική αξιολόγηση κινδύνου έχει γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτή η αξιολόγηση δεν ε, όρισε τα ωφέλη έναντι του κόστους. Βασίστηκε σε ένα διαφορετικό σχέδιο της ε, οδηγίας σε ό,τι αφορά λοιπόν τις προδιαγραφές της οδηγίας, την έκθεση, το κόστος βασίστηκε σε διάφορα σε διαφορετικές απαιτήσεις. Αυτό είναι σημαντικό για την συζήτηση που διεξάγεται στην παρούσα φάση σε ό,τι αφορά τις αρχικές, τον αρχικό υπολογισμό του και πάλι έγινε το σχόλιο ότι ήταν περιορισμένα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις μελέτες που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε πολλές λεπτομέρειες για το κόστος, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς από πού προήλθαν αυτές οι λεπτομέρειες. Και τέλος βλέπετε τον αριθμό των επιχειρήσεων που επηρεάζονται. Νομίζω ότι η Επιτροπή ε, δεν εκτίμησε σωστά τον αριθμό των επιχειρήσεων που επηρεάζονται. Νομίζω ότι έγιναν μεγάλα λάθη στο σημείο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εξήγησε τις κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα εργασίας. Δεν θα ήθελα να επισέλθω και εγώ σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να κοιτάξουμε εδώ είναι οι οριακές τιμές, η ρήτρα ευελιξίας και θα έλεγα και η ιατρική εποπτεία. Από πλευράς λοιπόν της ε, βιομηχανίας, της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Καλωσορίζουμε το κείμενο που έχει ήδη δημοσιευθεί που μιλάει για τα διάφορα είδη τιμών έκθεσης σε ό,τι αφορά την ευελιξία και πάλι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα σε κάποιους βιομηχανικούς κλάδους όπου ενδεχομένως τα όρια έκθεσης μπορεί να υπερβληθούν. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι και με δυνατότητα απόδειξη κίνδυνοι υγείας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη ευελιξίας για το θέμα της ιατρικής εποπτείας τώρα και παρακολούθησης. Το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ισχύον πρωτόκολλο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γιατροί για να μετρήσουν τη δοσολογία, την ποσότητα ακτινοβολία στο σώμα ενός εργαζόμενου. Άρα, οι ανεπιθύμητες παρενέργειες τις οποίες συζήτησα, ε, ανέφερα, Οι τιμέ λοιπόν οι οριακές μπορούν να υπερβληθούν για, πολλούς, για πολλές κοινέ διαδικασίες. Για παράδειγμα, στο, σε εφαρμογέ για τον διάστημα, διαστημική βιομηχανία. όπου μπορεί να περιπληθούν όχι μόνο τα όρια δράσης, αλλά και τα όρια έκθεσης. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αν δεν υπάρχουν επιθυμητές ενέργειες ή αν, είναι, ε, υπάρχει δυνατότητα αναστραφής τους, θα έπρεπε να αποκορευτούν αυτές οι διαδικασίες. Τελευταία διαφάνεια. Ποια κριτήρια θα έπρεπε να λάβει υπόψη η Επιτροπή αυτή για να κρίνει την ε, σημερινή πρόταση. Καταρχάς, να δούμε κατά πόσον η ομάδα εργασίας έχει ε, ανταπεξέλθει στις αρχές τις βασικές. Νομίζω ότι ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και ρεαλιστική δυνατότητα εφαρμογής των τιμών που ορίζονται κάποιες διαδικασίες ενδεχομένω να αποκλειστούν από το τομέα εφαρμογής της οδηγίας. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ποιο είναι το κόστος που το ξέρουμε και θα πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι τα ωφέλη. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα είναι αν υπάρχουν όντως βλάβες και κατά πόσον είναι δυνατόν αυτές οι βλάβες να αναστραφούν. Θα πρέπει τα μέτρα να είναι αναλογικά, θα πρέπει να είναι ευέλικτα, θα πρέπει να είναι κατανοητά στους εργοδότες και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής τους. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν η διαπραγμάτευση ήταν, θα είναι εύκολη. Υπάρχει μια λίγο πολυπλοκότητα όσον αφορά και το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις. Η κυρία Ντελή, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, σημείωσα μία σύγχυση στον ορισμό των κινδύνων, γιατί από τη μία μιλάμε για ανεπιθύμητες επιπτώσεις για την υγεία και για την ασφάλεια και τα ψυχολογικά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την ασφάλεια. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν, να σας ρωτήσω λοιπόν, ε, τι, γίνεται με αυτή τη σύγχυση, υπάρχει αυτή η διάκριση. Έπειτα, τι θεωρείτε όσον αφορά διαφορά μεταξύ ε, τιμών ε, αναφοράς και τιμών ε, δράσης. Επίσης, θα ήθελα να φέρω την έκθεση των εργαζομένων σε διαφόρους τύπους κυμάτων είναι λογικό κατά την άποψή σε αυτοί οι διάφοροι τύποι κυμάτων να τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης. Για παράδειγμα, η προειδοποίηση για τις χαμηλές συχνότητες. Δεν αναφέρθηκαν οι επιπτώσεις που συνδέονται με την επανάληψη, με την επαναλαμβόμενη έκθεση που έχουν μέσω ή μακροπρόθεσμα κάποιες πλευρές επιπτώσεις. Επίσης, όσον αφορά τις αποκλήσεις, τις παρεκκλήσεις, ιδιαιτέρως για το MRI, τι πιστεύετε εδώ. Δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ του συνήθους εξοπλισμού και αυτού που χρησιμοποιείται για, την έρευνα, όπου η υπέρβαση των ωριακών τιμών θα μπορούσε να θεωρηθεί λογική. Ε, βεβαίως, ε, υπό την προπόθεση θα λαμβάνονται επιπλέον ε, μέτρα ασφαλείας, εφόσον υπάρχει και αύξηση του επίπεδου κινδύνου. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τέσσερις εμπειρογνώμονες. Θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπαν. Επίσης το περιεχόμενο αυτού του φυλαδίου. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερος για το MRI. Και θα θυμάστε ότι η επιτροπή αυτή, στην επιτροπή είχαν μιλήσει δύο εμπειρογνώμονες αμέσω μετά την έκθεση της οδηγίας του 2004. Ήταν ιατροί ειδικοί από νοσοκομεία του Λονδίνου και είπαν ότι τα όρια που τίθενται σε αυτή την οδηγία είναι πολύ χαμηλά και και είπαν ότι αν είχαν εφαρμοστεί θα σταματούσαν τελείω τα ε, μηχανήματα μαγνητικής απεικόνηση. Επίσης είπαν ότι δεν υπήρχαν πουθενά σε κανένα νοσοκομείο στατιστικά στοιχεία για τα οποία προέκυπταν ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας είχαν υποστεί βλάβες λόγω των μηχανημάτων MRI. Αυτό σκεφτόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, σκεφτόταν, όταν όρισε αυτά τα όρια. Και Καταλαβαίνω πλήρως ότι όταν εργάζεται κανείς σε τέτοια παιδεία μπορεί αυτό να οδηγήσει σε βλάβες και σε βλάβες των ιστών συγκεκριμένα λόγω υπερθέρμανσης. Αλλά όπως σας είπα, τα όρια είχαν τεθεί υπερβολικά χαμηλά και αν είχαν εφαρμοστεί θα είχε σταματήσει η χρήση των MRI. Πρόεδρε λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Άκουσα όλα όσα είπατε σήμερα το απόγευμα και πρόσεξα ποια ήταν τα μη δεσμευτικά τμήματα τη σύσταση. Θα μπορούσαν ε, να με διαβεβαιώσουν οι δύο εμπειρογνώμονε ότι θα είναι ικανοποιημένοι και θα θεωρούν και θα είναι αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί η χρήση των MRI χωρί διακοπή. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα ζήτημα αυτό που συζητάμε τώρα ε, από τη μια μεριά πάρα πολύ τεχνικό και από την άλλη μεριά αγγίζει πάρα πολύ το θέμα της οικονομίας και το θέμα της εργασίας και βεβαίως ε, το θέμα της υγείας. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν αφορούν μόνο το MRI, MRI ε, αλλά εκ των πραγμάτων εστιάζουμε εκεί. Ε, κάνουμε μία προσπάθεια, αυτό τουλάχιστον έχω εγώ στο μυαλό μου, σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε μέσα σε αυτή την Επιτροπή, να μπορέσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Ασφάλεια για αυτούς που χειρίζονται τα μηχανήματα, ασφάλεια για αυτούς που εκτίθενται ως ασθενείς για παράδειγμα και ταυτοχρόνως ε, ασφάλεια εντός εισαγωγικών για τους εργοδότες, να το πω έτσι. Όταν λέω εργοδότες δεν εννοώ μόνο τον ιδιωτικό τομέα, γιατί ένα δημόσιο νοσοκομείο ας πούμε το οποίο έχει μαγνητικό τομογράφο είναι εργοδότης των γιατρών. Άρα έχουμε και το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα να εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Αισθάνομαι ότι θα πρέπει να δούμε ε, όρια και διασφαλίσεις που να είναι μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στη ζωή. Ε, τα μηχανήματα καθώς εξελίσσονται αυξάνουν, το λέω με τα απλά λόγια ενός ανθρώπου που δεν είναι ειδικό ε, και δεν χρησιμοποιεί ορολογία, αλλά οι ειδικοί μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά τι εννοώ, ε, αυξάνονται οι κίνδυνοι. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και εμείς την ασφάλεια. Και όλα αυτά με το λιγότερο δυνατό κόστος. Αλλά Τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω ότι το κόστος έχει δύο όψεις. Υπάρχει το οικονομικό κόστος και υπάρχει το κόστος στην επιβάρυνση της ανθρώπινης ζωής. Θα πρέπει να τα δούμε σε μια ισορροπία. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και η σημερινή ακρόαση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της καλής συναδέλφου, της κυρίας Αρτιέ, όπως ήταν πολύ χρήσιμες και οι άλλες δύο διαβουλεύσεις που έγιναν. Νομίζω ότι έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε ακόμη και θα πρέπει να έχουμε, αν μη τι άλλο, μεταξύ μας όλοι οι φορείς που εμπλεκόμεθα σε αυτή την υπόθεση, καλή διάθεση και καθαρή διάθεση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κυρία Μωρά. Ωραία, λοιπόν, άκουσα καλά τους τρεις ε, παρεμβαίνοντες μετά την Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι ο κύριος Σαπίρ υπήρξε ιδιαίτερος ακριβής όσον αφορά το γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καλυφθούν. Ε, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει κατά την άποψή σας να συμπεριληφθούν όλα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ή θεωρείτε ότι μπορούν να υπάρξουν εθνικές οδηγίες εφαρμογής. Εγώ έχω μία ερώτηση για την Επιτροπή. Αφού μου λένε ότι το Συμβούλιο πήρε το κείμενο και τροποποίησε τόσο τη δομή όσο και το περιεχόμενο του κειμένου. Ε, πώς ε, εσείς αντιμετωπίζετε αυτή την ανασύνθεση του κειμένου και μέρους του Συμβουλίου. Θεωρείτε ότι σε εκφράζει, θεωρείτε ότι συνιστά μια βελτίωση, θεωρείτε ότι υποεπίτευξη επίτευξη στόχοι έχουν ε, επιτευθεί. δεν ξέρω κατά πόσο όλοι μπόρεσαν μέχρι στιγμής να αναλύσουν τα αποτελέσματα ε, αυτού του ξεπλήματος. Λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο σε αντίστροφη σειρά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τον κύριο Βόλμαρ που μίλησε τελευταίος. Ως αν θεωρείτε βεβαίως ότι δεν έχετε κάτι να προσθέσετε. Sorry, I'm not, I'm not used to the process within this particular... Θέλετε να απαντήσω σε όλα τα σχόλια, γιατί δεν γνωρίζω τη διαδικασία που ακολουθείτε στην Επίτροπη την Επιτροπή. Είμαστε στο τέλος της ακρόασης και δεν ξέρουμε κατά πόσο θέλετε να απαντήσετε ή να αντιδράσετε σε όσα ελέγχθησαν από τα μέλη. Υπήρξε ένα ε, ερώτημα για τις ε, τιμές προσανατολισμού. Μπορώ να σας δώσω αυτές τις πληροφορίες τώρα ή μετά την ακρόαση σε σχέση με αυτές τις ε, τιμές, αν το κρίνετε σκόπιμο. If you're here, it's to give... Άμα θέλετε μπορείτε να μας δώσετε τώρα τις πληροφορίες. Εκτός αν χρειαστείτε μία ώρα. Εντάξει, οκ. Okay. τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ως προς τις τιμές προσανατολισμού. Αν η έκθεση είναι κάτω από το επίπεδο προσανατολισμού για χαμηλότερες συχνότητες δεν αναλαμβάνει καμία δράση γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους εργαζόμενους. Αν όμως η έκθεση είναι πάνω από τις τιμές προσανατολισμού για λόγους ασφάλειας, και αν έχει κρίσιμη εργασία, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να γνωρίζει κατά πόσο γίνονται υπερβάσεις. Εάν δηλαδή κάποιος έχει πονοκεφάλους ή ναυτίες λόγω συχνοτήτων, δεν θα θέλαμε να εργάζεται σε υψόμετρο. Και αυτό θα πρέπει να το ορίσει ο εργοδότης. Επίσης, ο εργοδότης θα πρέπει να προσδιορίσει κατά πόσο χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας, έτσι ώστε να μην υπερβούμε τα action values και θα πρέπει να μην υπερβούμε τα επίπεδα έκθεσης. Εάν οι οριακές τιμές δηλαδή τύχουν υπέρβασης, και εδώ μιλάμε για τη ρήτρα ευελιξίας, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να επαληθεύσει κατά πόσο οι εργαζόμενοι βρίσκονται υπό έλεγχο και δεν πλήττεται η υγεία τους. Ο κύριος Μάρκ Σαπίρ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις. Το πρώτο θέμα αφορά την υγεία και την ασφάλεια στις χαμηλές συχνότητες. Θα ήθελα να σας πω τι μου κάνει εντύπωση. Όταν μιλάμε για τις ΙΠΑ, για τα μαγνητικά πεδία βλέπουμε στατιστικές όπου βλέπουμε ότι αυξάνονται τα ατυχήματα διότι τα ε, μέταλλα προσελκύουν αυτές τις συχνότητες. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει ένας διαχωρισμός. Εγώ είχα ήδη πέσει η πτώση, εντάξει, ξέρουμε πώς ορίζεται, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή το συμβάν από τις απόρριες του συμβάντος. Δηλαδή, μας ε, ενδιαφέρει να ξέρουμε ότι, του χάρη, μπορεί να κρατήσει την ισορροπία του, ότι δεν θα πέσει, αλλά και τι θα γίνει μετά. Πιστεύουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί στα MRI ε, λένε στις ΕΠΑ ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων γιατί κανείς εξετάζει πολλούς ασθενείς και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι μία προσέγγιση των οριακών τιμών, η προσέγγιση αυτή των οριακών τιμών όπως έχει τώρα, δεν είναι σωστή. Μιλάμε, για, μιλάμε με υπεραπλουστεύσεις. γιατί θα πρέπει να ερμηνεύσουμε και αυτές τις ε, μετρήσεις in situ. Αυτό είναι το δύσκολο. Και για να απαντήσω στο τελευταίο σημείο, θα πρέπει να δούμε μέχρι πού θα εναρμονίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με το εθνικό. Ξέρουμε ότι οι οδηγίες απευθύνονται στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρουν τα μέσα για τη θέση σε εφαρμογή η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Έχετε έναν κατάλογο χωρών που δεν διαθέτουν νομοθεσία, ενώ άλλες ήδη διαθέτουν. Το να βρούμε μία σωστή ισορροπία είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό προσπάθησα να σας πω και πριν. Οι οριακές τιμές θα πρέπει να είναι σαφέστατες για να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε και να τις κατανοήσουμε και θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και η δοσομέτρηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην οδηγία για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις διάφορες ε, τεχνολογικές καταστάσεις. Θα ήθελα όμως να πω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ορίσουμε μία ομάδα εμπειρογνωμών για να παρακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και να δούμε πώς εξελίσσουν τα πράγματα, διότι στις, μαγνητικές, στις πυρηνικές μαγνητικές απεικονίσεις βλέπουμε ότι υπάρχει ε, διαφορετική, ε, διαφορετικές επιπτώσεις αν βρισκόμαστε στο 1,5, στο 5, στο 8 ή στο 11. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η επιτόπια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε αφηρημένα. Θα πρέπει να συνδέσουμε τη γενική συζήτηση με την ειδική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν τώρα για τη Business Europe, κυρία Ρεβέκα Σμιθ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα των αποκλήσεων κλπ. Νομίζω ότι θα ήταν προκειμένου να υπάρξει ευελιξία στην οδηγία. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όπως λέχθη όλοι οι τομεί ε, καλύπτονται από την οδηγία. Δεν μιλούμε λοιπόν για ειδικέ αποκλήσει εδώ, παρακλήσει εδώ, αλλά μιλούμε για αρισμένα στοιχεία περιορισμένη ευελιξία. Έχουμε την περίπτωση των MRI, που προφανώ είναι πολύ ξεκάθαρη και ιδιαίτερα σημαντική, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι ο μόνο τομέα ο οποίος επηρεάζεται αρνητικά τουλάχιστον από την παρούσα πρόταση και όπου θα υπάρξουν δυσκολίες ε, εφαρμογής των οριακών τιμών στην ε, παρούσα πρόταση. Από την άποψη της Business Europe ε, είμαστε μια ένωση εργοδοτών και θεωρούμε ότι αν η οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς, αυτό θα είναι προβληματικό. Ε, παρόλα Παρ' όλα αυτά, ε, ε Βεβαίω υπάρχει το θέμα ε, της τη εφαρμογή στον τομέα τη υγεία όσον αφορά το MRI, αλλά επίση και ορισμένε διαδικασίε συγκόλληση. Και αυτό λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η οδηγία έχει αρνητικέ επιπτώσει σε τέτοιου είδου διαδικασίες χρειάζεται μια ποσότητα ευελιξίας. Βεβαίω αυτό θα πρέπει να γίνεται κάπου από ελεγχόμενε προποθέσει και νομίζω ότι εδώ έγκυται το κλειδί τη υπόθεση. Είναι δύσκολο να δούμε αυτή τη στιγμή το πώ όλα αυτά θα εξελιχθούν, για παράδειγμα όσον αφορά τα ζητήματα του MRI, αλλά νομίζω ότι από τη δική μα άποψη ήδη έχουμε ως ε, βάση την οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια που υποχρεώνει τους εργοδότες να αναλάβουν ε, μελέτες εξολόγηση του κινδύνου για του εργαζόμενες και πιστεύω ότι κάθε είδους ευελιξία θα πρέπει να στηρίζεται από ειδικά μέτρα ελέγχου ή άλλα, για παράδειγμα, όπως υπόθηκε ήδη, να οργανώνεται η εργασία κατά τρόπο που, για παράδειγμα, να μην δουλεύει κανείς σε μεγάλο ύψος ε, αν κάποιος πάσει από ελέγχους. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κάποιου ε, πάση φύση πρακτικά μέτρα για να επιτρέπουν αυτού του είδο την ευελιξία. Θα ήθελα να επανέλθω στο σημείο το οποίο τέθηκε από, την, ε, από το συνάδελφο από την ETUC, όπου προφανώς υπάρχει διαφορά απόψεων όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ επιπτώσεων για την ασφάλεια και επιπτώσεων για την υγεία. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι μια διάκριση κλειδί εντός της οδηγίας. προφανώς η οδηγία θα πρέπει να προστατεύει αποτελεσματικά τους εργαζόμενους από τις επιπτώσεις τόσο στην υγεία όσο και στην ασφάλεια. Αλλά θεωρώ ότι είναι διαφορετικά διακριτά πράγματα. Πρώτον, η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε ένα υψηλό επίπεδο μπορεί να έχει μια επίπτωση στην υγεία των εργαζομένων. Αλλά είναι διαφορετικό εάν έχει στην ασφάλεια των εργαζομένων. Βεβαίως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θέματα όπως είναι τα ατυχήματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των εργαζομένων, αλλά ε, είναι μόνο μια δυνατότητα, ένα ενδεχόμενο να οδηγήσει σε τέτοιου είδους ατυχήματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η διάκριση είναι τέλος χρήσιμη από τη δική μας οπτική γωνία, όπως είπα προηγουμένως, και επίσης ε, ταιριάζει το, την, το λοιπό κορμό της οδηγίας όσον αφορά τη διαφοροποίηση μέτρων εκ μέρους των εργοδοτών όσον αφορά τα μέτρα υγείας και τα μέτρα ασφαλείας. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Σερμιγιόν εκ μέρους της Επιτροπής. Θα ξεκινήσω απαντώντας στην ερώτηση της κυρίας ε, Προέδρου και θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο για τα λοιπά ερωτήματα. Ε, αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία εξέτασης των συμβιβασμών που παρουσίασε η Προεδρία. Αυτή είναι μια πρώτη λοιπόν εντύπωση σε σχέση με αυτή την πρόταση παρά τις ε, αλλαγές όσον αφορά ορισμένα άρθρα, επί της ουσίας θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή δεν θέτει ένα αφιβόλο τους ουσιαστικούς σκοπούς της Επιτροπής με την πρόταση αυτή. Δηλαδή, θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της οδηγίας, συνεπώς τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων έναντι της ε, έκθεσης σε κινδύνους, και το κάνουμε μέσω της ε, διατύπωσης κάποιων ε, ε, αξιών, κάποιων κριτηρίων και εισάγουμε και την ευελιξία που επιτρέπει την εφαρμογή της οδηγίας σε ολόκληρη την βιομηχανία, στα νοσοκομεία καθώς και το στρατό και τέλος θέλουμε να προβλέψουμε μια προσαρμογή αυτών των τιμών ούτως ώστε ε, στην περίπτωση που η τεχνολογική εξέλιξη απαιτήσει νέε τιμέ τη θέσπιση νέων τιμών. Αυτή η στόχη δεν να αφιβόλου από την πρόταση. Ε, βεβαίως υπάρχουν ορισμένες πτυχές, όπου ορισμένες προτάσεις ε, παρεκκλίνουν από την πρόταση της Επιτροπής και ήδη αναφέρθηκαν οι υποχρεώσεις για την επιχείρηση όσον αφορά την ιατρική επίβλεψη και θεωρώ ότι αυτές οι υποχρεώσεις αλλαγιστοποιούνται στην πρόταση συμβιβασμού Επίσης υπάρχει μια ίσως υπερβολική απλούστευση όσον αφορά τις τιμές προσανατολισμού και τις τιμές δράσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιες δυσκολίες εφαρμογής στο βιομηχανικό τομέα ηλεκτρισμού και ε, επίσης καταργήθηκε ο κατάλογος του εξοπλισμού που μέχρι τώρα ήταν ένας τρόπος όπου η Επιτροπή είχε φανταστεί ότι μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά ενδεχομένω θα υπάρξει δυνατότητα να αντικαταστήσει αυτό ο κατάλογος του εξοπλισμού στην οδηγία από άλλα μέσα επιδιώκοντας, ε, εκπληρώνοντας τον ίδιο σκοπό. Ευχαριστώ κύριε Σίλβα. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με την ε, ονοματολογία, δηλαδή τα safety effects και τα health effects, τις επιπτώσεις για, επί της ασφάλειας και επί της υγείας. Μιλάμε για επίπεδα αναφοράς που στην οδηγία του 2004 μεταφέρονται ως action values, δηλαδή ως αξίες δράσης. Και υπάρχουν και οι οριακές τιμές έκθεσης. Αλλάξαμε την ονοματολογία τέσσερις φορές και εδώ στις νέες, στις νέες συστάσεις, όταν μιλάμε για χαμηλές συχνότητες, γιατί για τις υψηλές συχνότητες δεν άλλαξε τίποτα, από 0 έως 100 kHz έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι η ΚΝΙΡ έκανε μία διάκριση. Η ΚΝΙΡΠ. Δηλαδή μιλήσαμε για το κεντρικό νευρικό σύστημα και το περιφερειακό νευρικό σύστημα. Με συγχωρείτε, το αντίστροφο λέει ο μιλητής. Δηλαδή για το περιφερειακό νευρικό σύστημα που είναι το σώμα και το κεντρικό νευρικό σύστημα που είναι ο εγκέφαλος. Εάν λοιπόν κοιτάξετε στην ΙΚΝΙΡΠ έχετε δύο σειρές οριακών τιμών. Όμως οι τιμές αναφοράς που είναι τιμές δράσης αναφέρονται σε μία καμπύλη και εκεί καινοτομήσαμε με βάση τα στοιχεία που βρίσκουμε στην, που βρίσκουμε στην ε, τεκμηρίωση. Δηλαδή φτάσαμε σε μία δεύτερη καμπύλη και γι' αυτό μιλήσαμε για orientation values, ε, δηλαδή για τιμή προσανατολισμού και τιμή δράσης. Action values. Γιατί όπως ξέρετε κύριε Σαπίρ, το ανθρώπινο σώμα είναι λίγο πιο περίπλοκο από το κεφάλι και το σώμα ξεχωριστά. Και γι' αυτό μιλάμε για safety effects και health effects. Τα safety effects, δηλαδή οι οριακές τιμές για τις επιπτώσεις της ασφάλειας, σχετίζονται με τη φωσφίνη, δηλαδή ε, τα μικρά σαμιγάκια που βλέπουμε στα μάτια, και δεν θεωρούμε ότι είναι του ίδιου επίπεδου με άλλες επιπτώσεις που βρίσκουν πιο ψηλά στην ιεράρχηση. Έτσι μας λέει και η ΚΝΙΡΠ και έτσι βλέπουμε, βάζουμε σε μια προοπτική τις διάφορες επιπτώσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μια αναλογικότητα και ευελιξία όπως ζητούν οι επιχειρήσεις. Και επιμένω ότι η Κομισιόν κράτησε ένα υψηλό επίπεδο, ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των εργαζομένων. Είναι ένα περίπλοκο σύστημα, το αναγνωρίζω, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, αλλά τη στιγμή που υπάρχουν οδηγίες χρήσης θα είναι εύκολο εφάρμοστο. Ως, το, ως προς το MRI, τη μαγνητική απεικόνηση, γιατί μετά το 2004 είχαμε ακτινολόγους οι οποίοι μας είπαν ότι με την οδηγία του 2004 και τις οριακές τιμές της εποχής δεν μπορούσαν πια να εργαστούν. Μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή εργάστηκε επίπονα και ήρθε σε επαφή με τους κατασκευαστές και με τους ακτινολόγους και τις ενώσεις των ασθενός, το λεγόμενο Alliance for MRI και στις δύο ομάδες εργασίας και ιδιαίτερα στους ακτινολόγους βλέπουμε ότι είναι οι ίδιοι στους οποίους αναφέρεται και ο συνάδελφος και γνωρίζει πολύ καλά. Κάναμε πολλά λοιπόν σε επίπεδο Επιτροπής ποσοστοποιήσαμε, μάλλον είδαμε ποσοτικά το φαινόμενο, διότι υπάρχουν διάφορες, υπάρχουν διαβαθμίσεις και μετά από μία μελέτη του 2008 της Κομισιόν μιλήσαμε, εάν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν 10 εκατομμύρια υποθέσεις στα 27 κράτη-μέλη για τη μαγνητική ε, απεικόνηση, δεν υπάρχουν προβλήματα στις περισσότερες ε, εξετάσεις ρουτίνας. Αλλά σε 10-15% των περιπτώσεων θα πρέπει να αλλάξουμε κάπως τον τρόπο εργασίας. Και υπάρχει ένα 5-6-7% υποθέσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μιλάμε για πληθώρα υποθέσεων, γιατί μιλάμε για νέες οριακές τιμές σε σχέση με το 2004. Θα πρέπει να σταματήσουμε τις ε, μαγνητικές απεικονίσεις εξαιτίας αυτού. Βεβαίως όχι. Φυσικά θα πρέπει να προστατεύσουμε ιατρικά τους ε, ε, ανθρώπους του επαγγέλματος. Και τους είπαμε ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση αν εργαστούμε από κοινού για να αναπτύξουμε ενισχυμένα μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα που να έχουν επιπτώσεις ως προς τις αίθουσες μαγνητικής απεικόνησης, τον τρόπο εργασίας, τον κρατάει κανείς αποστάσεις, δηλαδή να ενημερώνεται καλύτερα ο εργαζόμενος και να έχει ένα εγχειρίδιο ας πούμε λύσεων συμφώνησαν. Για να απαντήσω στον κύριο Κλαπ, κατά πόσο με το παρόν σύστημα όσοι ασχολούνται με τη μαγνητική απεικόνηση είναι ικανοποιημένοι και η απάντηση είναι ναι. Εάν πάτε στον ιστότοπο της Alliance for MRI ή στους κατασκευαστές βλέπετε ότι συμβαδίζουν απολύτως με αυτό που προτείνουμε στο κείμενο και στο παράρτημα. Μπορούμε να μην συμφωνούμε 100% αλλά μπορώ να σας πω ότι όσο αφορά τη θέληση να βρούμε μια λύση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και να απτύξουμε αυτές τις τεχνικές για τους ασθενούς, μπορώ να σας πω ότι καταβάλαμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία εισηγήτρια, θέλετε να ολοκληρώσετε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή το σύνολο των εμπειρογνωμόνων σήμερα και καθώς και τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τους συναδέλφους. Νομίζω ότι μπορούμε από όλα αυτά να συναναγάγουμε μία γενική γραμμή συνένεσης όσον αφορά το εξή. Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι ε, δουλεύουν ε, με ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υγεία τους και η ασφάλειά τους. Ε, θεωρούμε ότι αυτό είναι απολύτως ε, θεμελιώδε. Δεν θα πρέπει συνεπώς ε, να αποκλείονται κάποιοι κλάδοι, κάποιοι τομεί εργασίε, αλλά θα πρέπει να γίνονται προσαρμογές σε συνάρτηση των ειδικών αναγκών και έστω και αν είμαστε πολλοί που έχουμε σκύψει στα προβλήματα που συνδέονται με τον τομέα της υγείας, ο τομέας του, αναφέρθηκε και ο στρατός, η άμυνα. Όλοι λοιπόν οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατοχυρώνονται, αλλά να υπάρχει μια ευελιξία στην προσαρμογή. Δεύτερο σημείο που τονίστηκε είναι το εξή. Μία, θα πρέπει να υπάρχει οδηγία που να είναι λειτουργική και εφαρμόσιμη. Και νομίζω ότι επί του σημείου αυτού υπάρχει γενική βούληση. Τρίτον, βεβαίως, η γενική κινητοποίηση ούτω ώστε η τεχνολογία των MRI και βεβαίως ο καθένας σκέφτεται την υγεία του γιατί όλοι είμαστε δυνητικά τουλάχιστον ασθενεί χρήστε του MRI η χρήση του MRI θα πρέπει να είναι απολύτω συμβατή με τη νέα μας οδηγία και ε, μένω στο να διευκρινίσω στον συνάδελφο κύριο Κλάρκ ότι χθε μαζί με τους συναδέλφους ε, εισηγητές, τη Σιλβάνα, τον Καρίν κλπ. Ε, ακούσαμε ε, την Alliance για τα MRI και μπορέσαμε να επαληθεύσουμε ακριβώς αυτό το οποίο διευκρίνησε προηγουμένως ο κ. Σερμπιγιό, δηλαδή τη συμβατότητα μεταξύ των δικών σας και των δικών μας ανησυχιών και φυσικά την ε, μελλοντική δυνητική χρήση του MRI. Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω ένα πράγμα, δηλαδή στην ε, δική μας οδηγία βλέπουμε και αυτό υπόθηκε ήδη το γεγονός ότι οι συσκευές στα μηχανήματα εξελίσσονται ραχδαία. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση όσον αφορά αυτές τις εξελίξεις. Ε, δεν μιλήσαμε, αλλά θα το ψάξουμε με τους συναδέλφους, υποθέτω, το ζήτημα του περιβάλλοντος του μηχανήματος. Υπάρχει το μηχάνημα και το περιβάλλον του. Το ίδιο το περιβάλλον του μηχανήματος, του, της συσκευής του εξοπλισμού, ε, είναι, ε, είναι ήδη είναι περιβάλλον ασφαλείας. Δηλαδή, ο εργαζόμενος, ο χρήστης, δεν ε, δουλεύει πάνω στο, μηχάνημα. Αλλά υπάρχει ακριβώς και το περιβάλλον. Δεύτερο σημείο, σε ορισμένες ε, περιπτώσεις ε, ε, ενισχυμένων κανόνων, βεβαίως η διατύπωση πρακτικών κανόνων για να πλουστευτεί και το έργο των επιχειρήσεων, αναφέρθηκε από πολλούς εμπειρογνώμονες στο θέμα αυτό, που τόνισαν ακριβώς την ανάγκη αυτός ο κανονισμός να είναι εφαρμοστέος, άρα εύληπτος, να μην προορίζεται απλώς και μόνο σε τεχνικούς αλλά ε, και από τους κατασκευαστές, από τους αλλά και από τους τεχνικούς στο ίδιο το εργασικό περιβάλλον. Επίσης θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με ένα σημείο στο οποίο επέμεινε η Σιλβάνα Ράπτη, δηλαδή ότι ε, θίγονται πολλοί τομεί και ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικό τομέας ε, άπτονται αυτών των ζητημάτων. Και βεβαίως υπάρχει μια οικονομική εφαρμογή και ε, σημαντικότατες οικονομικές επιπτώσεις ε, σε σχέση ακριβώς με τις αποφάσεις που θα λάβουμε. Και αυτό ισχύει τόσο για τον εξοπλισμό, όσο και για την εξέλιξη ακριβώς όλου αυτού του εξοπλισμού. Αλλά επίσης έχει και μια επίπτωση στις δαπάνες το κόστος υγείας. Εγώ ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό θα προσπαθήσω να προτείνω κάποιες τροπολογίες στο κείμενο της Επιτροπής ε, με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ε, αποτελεσματικότητα, δηλαδή λαμβάνοντας ε, υπόψη και τα όσα είπαμε εδώ και θα ήθελα να προσθέσω την κυρία Λιν, η οποία δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σήμερα εδώ. Είναι πολύ σύμφωνη με αυτή τη γραμμή σκέψης και ε, τονίζει ιδιαίτερα τους κινδύνους για τις, έγκυες, που εργάζονται, είναι υποχρεωμένες να εργαστούν σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και που θα πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερως. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Άρα ολοκληρώσαμε ή όχι. Σιλβάνα. Μπορώ να έχω το λόγο για λίγα δευτερόλεπτα. Από ότι ε, βάζοντας στο διαδίκτυο το MRI για το οποίο τόση ώρα κουβεντιάζουμε, όλοι θεωρούμε ότι μιλάμε μόνο για την, το Magnetic Resonance Imaging. Ε, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και κάτι άλλο που αντιστοιχεί στο MRI, το Mental Research Institute. Απλώς να το έχουμε στα υπόψη, για να βάλουμε λίγο χιούμορ μέσα στην κουβέντα μας. Bon. Bon. Mais pas Λοιπόν, δεν θα ξανά ανοίξουμε τη συζήτηση. Ήταν μια διευκρίνηση. Λοιπόν, επόμενο βήμα, η παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Μόρα στη συνεδρίασή μας στις 21ης και 22ης Δευτέρας. Ε, τελειώσαμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, παρατηρητές, τους βουλευτές και τους συνεργάτες τους. Ε, όσοι δεν είναι συντονιστές, παρακαλώ να φύγουν από την αίθουσα και ευχαριστώ και πάλι τους προσκεκλημένους μας που μας έδωσαν τα φώτα τους.